May I ask you take your seat so we can start. I would... Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, ας ε, θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνάμε απευθεία στο σημείο υπαριθμών 3. Ε, έχουμε τον νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο κύριο Ντράγκη, ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, πρόεδρο του κύριο Ντράγκη. Είναι ο δεύτερος νομισματικός διάλογος του 2019. Είναι ο πρώτος αυτή της ε, θητείας και βεβαίως και ο δικός μου πρώτος διάλογος με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Είναι βέβαια η τελευταία παρουσία εδώ του κυρίου Ντράγκη. Σίγουρα αυτό που ε, μας αποσχολεί περισσότερο είναι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να είναι χαμηλότερη από τον τελευταίο διάλογο. Ε, το ΑΕΠ ε, από 0,4% στο πρώτο εξάμεινο αυτού του έτους μειώθηκε σε 0,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο αυτού του έτους. Ενώ αντέχει η εσωτερική ζήτηση. Ε, παρόλα αυτά, λόγω των ε, διαφόρων γεωπολιτικών ε, παραγόντων, διαπιστώνουμε ότι οι γεωπολιτικοί αυτοί παράγοντες πιέζουν τον μεταποιητικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν κίνδυνοι που επίσης έχουν επηρεάσει την δυναμική εξέλιξη των τιμών. Υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά την εξέλιξη της, του πληθωρισμού με βάση το στόχο των μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Κατόπιν τούτου, πριν από 10 ημέρε, το Συμβούλιο της ΕΚΤ ανέφερε και ανακοίνωσε ένα πακέτο συμπληρωματικών μέτρων με στόχο να προσφερθούν οικονομικά κίνητρα. Και πιστεύω ότι ο κύριο Ντράγκη θα αναφερθεί περισσότερο σε αυτά στην εισαγωγική του παρέμβαση. Επίση, οι συντονιστέ τη ΕΚΟΝ επέλεξαν άλλα δύο θέματα για συζήτηση. Το πρώτο θέμα αφορά του παγκόσμιου ε, διαρθρωτικού παράγοντε. Ε, που επηρεάζουν ε, την μείωση τη δυναμική πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και γενικότερα. Και δεύτερον, τη στρατηγική που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Το δεύτερο, οι καινοτομίε υπό την Προεδρία του κυρίου Ντράγκη στο νομισματικό τομέα ε, και οι προκλήσει αυτά είναι εκείνα που μα απασχολούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο Εμεί ε, κάναμε μια προκατακτική εργασία. Μπορείτε να βρείτε σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα του αυτό βέβαια που μας ενδιαφέρει είναι και η άποψη της ΕΚΤ. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτός είναι ο τελευταίος νομισματικός διάλογος με τον κύριο Ντράγκη. Σήμερα οι βουλευτές που βλέπετε είναι η τρίτη επιτροπή ΕΚΟΝ στην οποία ε, έρχεστε να μιλήσετε μετά τον, την 7η και την 8η κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για τις επικοδομητικές σχέσεις που είχαμε τα τελευταία 8 χρόνια. Ήρθατε εδώ πάνω από 30 φορές ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και απαντήσατε σε πάνω από 600 ερωτήσεις. Η ΕΚΤ είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ επηρεάζουν τα μάλα, τις ευρωπαϊκές εταιρείε και τους ευρωπαίους πολίτες. Και με σίγουρα συμφωνείτε μαζί μου, ότι ο νομισματικός διάλογος ήταν και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη λογοδοσία ε, και ε, την διαφάνεια στην ΕΚΤ. Σας εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον και επιπλέον, επειδή μιλάμε για την αμοιβαία εκτίμηση, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω και ένα δώρο. Αυτό τον, τον ασημένιο δίσκο είναι εκ μέρους ε, όλων των μελών της ΕΚΟΝ, εκτός από την πολιτική ομάδα ID, Identity and Democracy.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 Uh, Πριν λοιπόν ε, δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ντράγκη, άκουσα ότι υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές ε, που θα ήθελα να συγκεντρωθούμε στην πρώτη σειρά για να βγάλουμε μια φωτογραφία. Καλύτερα λοιπόν να το κάνουμε τώρα και όχι αργότερα, που σημαίνει αν θέλετε να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Okay. Λοιπόν, ας επανέλθουμε στη δουλειά μας. Ε, κύριε Ντράγκη, έχετε το λόγο. Ε, thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα πάντα. Πριν ε, μπω στην εισαγωγική μου παρουσίαση, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, Θέλω πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ όλους για την ε, εκλογή σας. Και εσάς, κυρία Πρόεδρε, που οριστήκατε πρόσφατα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής αυτής Επιτροπής. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας, αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία. Και πριν ε, λήξει η δικιά μου θητεία, ω επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νομιμότητα στην οποία αναφερθήκατε και η ανεξαρτησία τη ΕΚΤ είναι πράγματα τα οποία γράφονται στι ίδιε τι συνθήκε και βασίζονται ακριβώ στη δικιά μα λογοθεσία. Και οι συνθήκε έχουν ε, επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα πάρα πολύ βασικό ρόλο, δηλαδή ότι λογοδοτεί η ΕΚΤ σε εσά. Η δικιά σα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, συνεπώ, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στη δικιά μου τη θητεία ε, θεωρώ ότι υποφελήθηκα πάρα πολύ από τις συναντήσεις που είχα μαζί σας. Όταν για πρώτη φορά ήρθα εδώ ενώπιον της ε, κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής το Δεκέμβριο του 2011, είχαμε μπει σε ένα στάδιο αβεβαιότητας, οικονομικής αβεβαιότητας και ένα δεύτερο στάδιο ήθεσης που οδήγησε σε ένα μεγάλο αποπληθωρισμό. Και μερικές φορές είχαμε και υψηλούς ε, κινδύνους υπερβολικού αποπληθωρισμού. Η Ευρωζώνη βέβαια έφτασε εδώ που έφτασε έχοντας διανύσει μεγάλο δρόμο χάρη στην βοήθεια της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ανεργία ήταν 7,5% τον Ιούλιο, που ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανειλημμένα έχει δείξει ότι είναι έτοιμη και αποφασισμένη να φέρει ε, πλήρως πέρας τον ρόλο της και τον στόχο της που είναι η σταθερότητα των τιμών έτσι όπως αναφέρεται και στις συνθήκες. Και ακριβώς η ετοιμότητα αυτή και η αποφασιστικότητά μας ήταν βασικά στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και η κίνδυνη να μην πετύχουμε το στόχο μας. Έτσι λοιπόν, με την ίδια αποφασιστικότητα, πριν από δύο εβδομάδε, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αντιδράσει εξαιτία ε, τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθωρισμού, προκειμένου να μπορεί να πετύχει το στόχο τη. Και χαίρομαι που μπορώ να συζητήσω τι αποφάσει αυτέ μαζί σα σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ποιες είναι οι πρώτες εξελίξεις από την προηγούμενη φορά που ήρθε εδώ. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις αποφάσεις σχετικά με την νομισματική πολιτική που υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τις προοπτικές. Και όπως ζήτησε η δικιά σας Επιτροπή θα ολοκληρώσω ε, προσπαθώντας να καταλήξω σε κάποια μαθήματα από το παρελθόν όταν συζητάμε για τις πολιτικές αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες προκλήσεις. Από την τελευταία ακρόαση που είχα εδώ, νωρίτερα αυτή τη χρονιά η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη επιβρανθήθηκε ήπια, περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει νωρίτερα. Η πραγματική ανάπτυξη του ΕΠ τώρα θα είναι 1,1% από ό,τι φαίνεται το 2019, 0,6% λιγότερο από τον Δεκέμβριο του 2018 και 1,2% προβλέπεται για το 2020 και πάλι χαμηλότερα 0,5% από τις προβλέψεις που είχαμε το Δεκέμβριο. Αυτή η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην αδυναμία που έχουμε εξαιτία του διεθνούς εμπορίου και στις επιμένουσες αβεβαιότητες που έχουν να κάνουν με γεωπολιτικούς παράγοντες. Και οι παράγοντες αυτοί ε, βαραίνουν πολύ και έχουν πλήξει και τον κατασκευαστικό τομέα που είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε ευπάθειες. Χώρες βέβαια οι οποίες έχουν μεγάλους τέτοιους κατασκευαστικούς τομείς είναι περισσότερο ευάλωτες σε οτιδήποτε πλήξει τον οικονομικό κύκλο. Η Γερμανία για παράδειγμα έχει κατά 28% του ΕΠ αλλά 39% τον ε, κατασκευαστικό τομέα σε προστιθέμενη αξία. Η Γερμανία επίση σήμερα είναι μία από τι χώρε μέλη της Ευρωζώνη που επηρεάζεται περισσότερο από την επιβράδυνση αυτή. Και ενώ ο τομέας των υπηρεσιών εξακολουθεί να αντιστέκεται, ε, δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να αντιστέκεται σε δευτερογενείς συνέπειες οι αδυναμίες στον κατασκευαστικό τομέα εφόσον συνεχιστούν, τότε κινδυνεύουν και άλλοι τομεί της οικονομίας, να επηρεαστούν δηλαδή από την οικονομική αυτή επιβράδυνση. Κοιτώντα προ το μέλλον πάντω, τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε και διάφορε δείκτε, όπω νέε εξαγωγέ, δεν δείχνουν σήματα για ανάκαμψη σύντομα και οι κίνδυνοι όσον αφορά την ε, μεγένθηση παραμένουν καθοδικοί. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών ε, των αδυναμιών της Ευρωζώνης, οι προπτικές όσον αφορά τον πληθωρισμό είναι κάτω από τα επίπεδα τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕ. Ο ε, ο, συγνώμη, ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός, ενώ παραμένει αστάθεια σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα, τις τιμές των τροφίμων, για παράδειγμα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, ο πληθωρισμός παραμένει αδύναμος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις ε, στην μετακύληση των μέτρων μας στις τιμές. Επίσης, οι επιχειρήσεις απορροφούν το κόστος εργασίας και δεν τα μετακυλούν στους πελάτες. Συγχρόνως, οι δείκτες όσον αφορά τις προσδοκίες για τον προπολογισμό βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλο που ο αποπληθωρισμός, οι προπτικές αποπληθωρισμού παραμένουν χαμηλές, παρόλα αυτά μεσοπρόθεσμα οι τιμές είναι τέτοιες οι οποίες δεν είναι συνεπείς με τους δικούς μας στόχους για τον πληθωρισμό. Από την τελευταία κρόασή μου εδώ αναθεωρήσαμε προς τα κάτω τις προπτικές ε, πληθωρισμού για όλη την περίοδο προβολής. Πρώτα απ' όλα τον Μάρτιο του 2019 με τις προπτικές των εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο ε, με χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα και χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 1,2% το 2019, 1% το 2020 και 1,5% το 2021. Κάτι το οποίο είναι πολύ κάτω από τους στόχους του Δικητικού Συμβουλίου που είναι να είναι κοντά πολύ αλλά κάτω από το 2%. Συνεπώ, όταν το Δικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε πριν από δύο εβδομάδε, είχε να αντιμετωπίσει μια ε, επιταχυνόμενη επιβράδυνση περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει κατά το παρελθόν. Επίμονη προς ε, τα κάτω όσον αφορά τις προπτικές και μη επιπλέον καθυστέρηση στη σύγκληση του πληθωρισμού προς τον στόχο μας. Μια ισχυρή νομισματική πολιτική λοιπόν ήταν αναγκαία. Για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας, αποφασίσαμε λοιπόν για ένα συνολικό πακέτο μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα πλησιάσει το στόχο μας και μάλιστα με ένα συνεπή τρόπο. Μειώσαμε λοιπόν το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων από το 0, ε, ε, μείον 0,4% στο μείον 0,5%. Το επιτόκιο αυτό μας ε, βοηθάει να ενισχύσουμε τα επιτόκια όπως θέλουμε και να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για διαφόρων ειδών δάνεια. Η μείωση των, ε, ε, του επιτοκίου διευκόλυνση αποδοχή καταθέσεων είναι κάτι το οποίο βοηθάει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσει. Τα αρνητικά επιτόκια επίσης ενθαρρύνουν τις τράπεζες να δανείζουν στην πραγματική οικονομία αντί να επιμένουν στην ρευστότητα και έτσι υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία του χαρτοφυλακίου και στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ενεργητικού. Τώρα οι επιπτώσεις της μείωσης αυτής ενισχύονται και από τις κατευθύνσεις μας στην νομισματική μας πολιτική για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, εμείς διευκρινίσαμε ότι αναμένουμε τα επιτόκια αυτά να παραμείνουν στο παρόν ή χαμηλότερο επίπεδο μέχρι να έχουμε δει ε, ότι θα παραμείνουν τα βασικά επιτόκια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα σημερινά σε χαμηλότερα επίπεδα, σε ό,τι επιστώσουμε ότι οι προοπτικέ για τον πληθωρισμό συγκλίνουν στεναρά προ επίπεδο πλησίων σε επαρκή βαθμό κάτω από το 2%, εντό χρονικού ορίζοντα προβολή που εξετάζουμε και ότι η σύγκληση αυτή αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού. Αυτές λοιπόν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, δίνουν ένα σήμα όσον αφορά τις ε, προσδοκίες γιατί συνδέουν ε, την πολιτική μας στις προπτικές που υπάρχουν τις αποπληθωριστικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης είπε ότι θέλουμε να αυξηθεί ο πληθωρισμός σε ένα επίπεδο αρκετά κοντά στο 2% αλλά κάτω από το 2%. Και ισχύει αυτό που είπαμε και τον Ιούλιο στην συνάντησή μας νομισματικού διαλόγου, ότι δηλαδή οι τιμές του πληθωρισμού, έτσι όπως βλέπουμε σήμερα, είναι ε, προς τα κάτω και όχι συνεπής προς τους στόχους ε, της ΕΚΤ. Η νέα διατύπωση λοιπόν τώρα κατευθυντηρίων γραμμών αντικατοπτρίζει τις ε, προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και προσθέτουμε και ρήτρες ασφαλείας έτσι ώστε η τακτοποίηση του ρυθμού να ξεκινήσει μόνο όταν θα είναι όταν θα έχει ε, αρκετά ε, ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας. Και θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί πριν αρχίσουμε να ε, αυξάνουμε τα επιτόκια. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να ενισχύει τις προπτικές μας. Οι κατευθυντήριες μας γραμμές αυτές λοιπόν θέλουν να μας βοηθήσουν ε, σύντομα, μεσοπρόθεσμα, να διασφαλίσουμε ότι οι δημοσιονομικές ε, προπτικές είναι αντίστοιχες. Επιπλέον, διατηρώντας τα επιτόκια αυτά, αν χρειαστεί, πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να τα μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Αποφασίσαμε επίσης να συνεχίσουμε τις ε, επενδύσεις από τον Νοέμβριο και μετά να συνεχίσουμε την αγορά δηλαδή στοιχείων ενεργητικού και ότι αυτό θα το κάνουμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και να ξέρουμε ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Επιπλέον, επαναλάβαμε ότι σκοπεύουμε να επανεπενδύουμε πλήρω τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στα πλαίσια του προγράμματο αγορά ενεργητικού κατά τη λήξη του για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια και πάντω για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθήκων ρευστότητα και διευκολυντικού σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα τη νομισματική πολιτική. Επίσης, θα ενισχύσουμε τον διευκολυντικό χαρακτήρα της πολιτικής μας για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά βοηθούν να διατηρήσουμε τα μακροπρόθεσμα επιτόκια χαμηλά, γιατί αλλιώς θα υπήρξε άνοδος αυτόματα κατά την λήξη του χαρτοφυλακίου. Τέλος, οι καθαρές αγορές αυτές δείχνουν και τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο της σταθερότητας των τιμών, κάτι το οποίο επηρεάζει και τις προπτικές ε, πληθωρισμού. Επιπλέον στα μέτρα αυτά τα οποία ανέφερα μέχρι τώρα, αποφασίσαμε επίσης να μεταβάλουμε τους όρους διενέργειας τη νέα σειρά τριμηνίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότηση, το τίλτρο 3 κάτι το οποίο ανακοινώσαμε ήδη τον Ιούνιο. Έτσι οι τράπεζες μπορούν τώρα να έχουν ε, με χαμηλότερα ε, επιτόκια όταν πρόκειται για μεγαλύτερη λήξη. Έτσι η... θα γίνει ομαλά η μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής και θα στηριχτεί παρετέρω η διευκολυτική κατεύθυνση της πολιτικής μας. Τέλος, επίσης, ανακοινώσαμε και ένα σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών, στο πλαίσιο του οποίου μέρος της πλεονέζουσας ρευστότητας που διακρατούν οι τράπεζες θα εξαιρείται από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Έτσι θα υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε δύο αποτελέσματα. Από τη μία διατηρούνται τα κίνητρα για τις τράπεζες προκειμένου να ε, βοηθηθούν από την τόνωση, την οικονομική και συγχρόνως τα αρνητικά αποτελέσματα από τα αρνητικά επιτόπια περιορίζονται όσον αφορά τη συμπεριφορά των τραπεζών σε σχέση με την επιθυμία τους για κερδοσκοπία. Χρειάζονται βέβαια διευκολύνσεις για να υπάρξει μετακύληση της πολιτικής μας αυτής. Το νέο σύστημα των δύο βαθμίδων θα ε, διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα δανείζουν περισσότερο από ευρωπαϊκούς όρους τους πελάτες τους. Θα ενισχυθούν τα μέτρα αυτά και με ευρωπαϊκές ε, συνθήκες χρηματοδότησης επιχειρήσεων όπως επίσης θα ενισχυθούν και οι δαπάνες των οικοκυριών με μια νέα δυναμική και έτσι θα μπορέσουμε πιο εύκολα να πετύχουμε το στόχο μας. Συνολικά όσον αφορά τις προοπτικές, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει να έχει διευκολυντικό ρόλο για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Τα μέτρα που πήραμε την τελευταία φορά και η ετοιμότητά μας να προσφέρουμε μέτρα οικονομικής τόνωσης θα συνεχιστούν και θα είμαστε έτοιμοι στο να προσαρμόσουμε ό,τι μέτρα χρειάζεται για να πετύχουμε τις προπτικές μας. Τώρα τα συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα, τα οποία έχει οθετήσει την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν επιτυχή για να πετύχουμε την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού, ε, γιατί καταφέραμε να ενισχύσουμε την μετάβαση των πολιτικών μας στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βέβαια δεν λειτουργεί μέσα σε ένα κενό. Υπάρχουν και άλλες οικονομικές ε, πολιτικές οι οποίες παίζουν ρόλο. Και εδώ ε, θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι είχα πει την πρώτη φορά το 2011 δηλαδή που είχα έρθει σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Τότε οι μισές από τις αγωγικές μου παρατηρήσεις ήταν για την λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και έλεγα ότι χρειαζόντουσαν και άλλες ε, πολιτικές συγχρόνως. Συνεπώς, θα ολοκληρώσω τονίζοντας τι μαθήματα έχουμε πάρει από τα 8 αυτά χρόνια που ήμουν επικεφαλή στην ΕΚΤ και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προσεχείς ε, προκλήσεις. Όταν συγκρίνουμε πώς αντιμετώπισε η Ευρωζώνη την κρίση σε σχέση με άλλες ε, περιοχές του κόσμου, είναι σαφές ότι υπήρξε καλύτερο μείγμα ε, οικονομικών μέτρων χάρη σε μέτρα που υιοθέτησαν και στο δημοσιονομικό τομέα όπως και στο νομισματικό. Εμείς φυσικά και θέλουμε να πετύχουμε τον πληθωρισμό βάσει του στόχου μας και είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε για να το πετύχουμε αυτό. Χρειάζεται όμως ένα καλύτερο πολιτικό μείγμα. Χρειάζονται δηλαδή και δημοσιονομικές πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προληπτικά μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε ε, τους στόχους μας πιο γρήγορα και χωρίς παρενέργειες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ελέγχουμε, όπως ε, καταλαβαίνετε, τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η διευκολυντική μας προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μικρό και μάκρο πολιτικής για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό ακριβώς ε, προσπαθώ να κάνω και εγώ και προσπαθώ πάντα να κάνω πρέπει να κατανοήσουμε το γενικό ε, περιβάλλον ε, στα πλαίσια ε, των όσων έχουμε δει από το 2008 και μετά. Κοιτάσει αυτή βέβαια δεν αφορά μόνο την Ευρωζώνη, έχει να κάνει με διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι η μείωση της αύξησης στην παραγωγικότητα, που μας οδηγούν σε διαφορετικά μέτρα. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιονομική που να ενισχύει τα μέτρα που παίρνουμε στην νομισματική πολιτική. Και υπήρξε στο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφωνία για το ότι η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να βοηθήσει στα πλαίσια των χαμηλών οικονομικών προοπτικών και των κινδύνων που υπάρχουν. Οι χώρες οι οποίες έχουν περιθώρια θα πρέπει να δώσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα δημοσιονομικά. Ε, όσες ε, μπορούν ε, να ε, ενισχύσουν στα σημεία του κύκλου που μπορούν να το κάνουν, πρέπει να το κάνουν. Συγχρόνως, οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος ε, πρέπει να επιδιώξουν την άσκηση συνετών πολιτικών και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών για να πετύχουν τους στόχους. Άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν αντικυκλικές ε, καταστάσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αντίστοιχε δυσκολίες υπάρχουν και όταν συζητάμε και για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και για την ολοκλήρωση τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Πρέπει ε, να φροντίσουμε να πετύχουμε μια πραγματικά αυθεντική ε, Οικονομική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς θα καταστρέψουμε τόσα ήδη έχουμε καταφέρει με τη σκληρή δουλειά όλων και πάνω απ' όλα της δικιάς σας Επιτροπής. Όπως έχω πει και πριν από 8 χρόνια εδώ σε αυτή την Επιτροπή, πρέπει να δείξουμε το δρόμο για τις μελλοντικέ εξελίξεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και έτσι να πλαισιώσουμε τις προσδοκίες τόσο των οικονομικών αγορών όσο και των πολιτών μας. Και επιτρέψτε μου τώρα να πω κάτι ακόμα για το τελευταίο μάθημα που πήραμε. Ενώ η Ευρωζώνη δεν είχε ε, δημοσιονομική πολιτική απάντηση αντίστοιχη με αλλού, παρόλα αυτά μπορούμε κάλλιστα να τη συγκρίνουμε με τα μέτρα που πήρανε άλλες τράπεζες. Με την ανεξαρτησία της η ΕΚΤ μπόρεσε να προσαρμόσει την δικιά της απάντηση και τη λειτουργία της, διατηρώντας το βασικό της στοιχείο που είναι η ανεξαρτησία της. Και έτσι μπορέσαμε να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις και να αποδείξουμε ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρηθεί γιατί δέχεται πιέσεις από πολλές πλευρές. Όμω, αυτό που είναι εξίσου σημαντικό για μας είναι η λογοδοσία μας και η πρακτική λογοδοσία μας ε, πιστεύουμε ότι είναι κάτι που εξελίσσεται όπω υπενθύμησε και η πρόοδο ακριβώς επειδή Εξαιτία τη ε, κρίση, μα ζητήθηκε όλο και περισσότερο έλεγχο. Πάντα εκτίμησα την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δρά βάσει των όσων ζητούν οι πολίτε και με επικοδομητικό τρόπο να ζητά περισσότερες εξηγήσεις από εμά. Σας ευχαριστώ προσωπικά όλους και είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή κυρίως θα συνεχίσει το καλό έργο που έκανε μέχρι τώρα και με την επόμενη πρόοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, οι δράσεις μας θα είναι πιο ισχυρές και θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντράγκη. Περνάμε λοιπόν τώρα στις ε, ερωτήσεις. Έχω τον κατάλογο των ε, ερωτώντων. Ε, πέντε λεπτά λοιπόν για τον καθένα για ερώτηση και απάντηση. Ο κύριος Μάρκους Φέρμπερ, παρακαλώ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε και εσείς ε, κύριε Ντράκη να μιλήσω γερμανικά. Και ευθύς εξ αρχής να πω ότι εκ μέρους του ΕΛΚ σας ευχαριστώ θερμά. Τα Ιταλικά τα μιλώ σπανιότατα, γι' αυτό λοιπόν ε, προτιμώ να μιλήσω γερμανικά. Φαντάζομαι με ακούτε. Λοιπόν, εκ μέρους του ΕΛΚ σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία οκτώ χρόνια και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν αναλάβατε το αξίωμά σας ε, θυμάμαι την ακρόαση που είχαμε τότε οργανώσει και νομίζω ήταν απόλυτα σαφές ότι δεν θα ήταν εύκολη η περίοδος που θα ακολουθούσε και όλοι μας γνωρίζαμε τι έπρεπε να αποφασιστεί στα οκτώ επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε εδώ σε τακτά χωρικά διαστήματα και δικαιολογήσατε πάντα τις αποφάσεις σας. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στις νομισματικές αποφάσεις που πολίτησαν την προπροηγούμενη εβδομάδα, ε, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων, να ξαναξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Πολλές κεντρικές τράπεζες ε, στράφηκαν κατά ε, της επανέναρξης αυτού του προγράμματος. Αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό, γιατί υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα της εξαγοράς των ομολόγων λόγω των εξελίξεων λόγω του πληθωρισμού, κατά πόσον αυτό ήταν απαραίτητο. Και ρωτώ, ε, μέσα στο Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ, ε, γιατί αποφασίσατε για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, κυρίως έχοντας κατά νου ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το περιθώριο κινήσεων της κυρίας Λαγκάρτ, που πρόκειται να αναλάβει τα ενία της τράπεζας. Έχοντας κατά νου ότι ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη παρά την ιδιαίτερα χαλαρή πολιτική ε, δεν έχουν αλλάξει, τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λάβατε τα τελευταία χρόνια, γιατί τελικά δεν συνέβαλαν έτσι ώστε να αυξηθεί ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει περίπου στον επιδιωκόμενο στόχο του 2%. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κατ' ουσίαν ε, θέσατε δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί λάβαμε αυτές τις αποφάσεις και δεύτερον, κατά πόσον είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι αποφάσεις θα είναι αποτελεσματικές τη στιγμή που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι κάτω από το στόχο μας. Θα θυμάστε στην αρχή, στην εισαγωγική μου ομιλία, ε, είπα και επαναλαμβάνω το εξή. Το θέμα των, το νομισματικό εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Βλέπουμε ε, να βελτιώνονται κάποιες αγορές, ε, εντάξει όχι με την ίδια δυναμική. βλέπουμε η κατανάλωση να είναι λιγάκι περισμένη, να βελτιώνονται λιγάκι οι επενδύσεις, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, το ποσοστό ενεργείας είναι το χαμηλότερο από το 2008. Και αυτό λοιπόν μας καθιστά αισιόδοξου ότι κάποια στιγμή ο πληθωρισμός ε, θα φτάσει εκεί που τον θέλουμε. Ε, αν λοιπόν στρέψει κανείς το βλέμμα στο μέλλον, θα διαπιστώσει ότι τα, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώνονται σταθερά. Και αν πάμε πίσω στο 2018, τότε ε, κάποιοι διαφώνησαν με τις αποφάσεις τότε είχαμε πει ότι η προσωρινή αυτή ανάπτυξη οφείλεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες εξελίξεις. Και τότε μας είπαν ότι αυτές οι βραχυπρόθεσμες εξελίξεις θα διαρκέσουν λίγο περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Εν τω μεταξύ προέκυψε η γεωπολιτική ανασφάλεια, η οποία επέτεινε συγκεκριμένους παράγοντες σε συγκεκριμένες χώρες και κατόπιν η παροδική επιβράδυνση ε, που είναι κάτι που υπάρχει, αν το 17 που είχαμε υπερβολική ανάπτυξη, όλα αυτά οδήγησαν στο να έχουμε ε, μία μεγαλύτερη επιβράδυνση, μία κοιλιά αν θέλετε, σε αυτό τον δρόμο της ανάπτυξης που κράτησε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και ε, αυτό το περιμέναμε, το είχαμε εκφράσει πριν από 6-7 μήνες. Η έκτη λοιπόν έχει αναθεωρήσει πολλές φορές ε, τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και αυτός είναι ο πρώτος λόγος γιατί το Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αναλάβει δράση. Ο δεύτερος λόγος είναι οι προοπτικές ε, ε, του πληθωρισμού. Ε, το πρόγραμμα Juncker εκφράζει κάποιες σκέψεις για δραστηριοποίηση Παρόλα αυτά, εμείς ε, προβλέπουμε ποσοστό πληθωρισμού 1,5 μέχρι το 2021, που είναι και το τέλος των προβλέψεών μας. Αυτό το 1,5% είναι πολύ πιο κάτω από το στόχο μας. Άρα δηλαδή έπρεπε κάτι να κάνουμε και αν δεν κάναμε κάτι θα έπρεπε και πάλι να υποβαθμίσουμε τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις μας και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε συμβατοί με την εντολή που έχουμε λάβει που είναι σταθερότητα των τιμών. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση δεύτερη απάντηση είναι ε, και τότε γιατί συνεχίζετε να λάβετε, λαμβάνετε μετά στιγμή που αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Θα απαντήσω ως εξή. Θα επανέλθω σε αυτό εντός λίγο, αλλά ας πάμε λίγο πίσω ή δεν έχω χρόνο. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω για άλλο ένα λεπτό. Λοιπόν, Ας πάμε πίσω στο 2014 όταν για πρώτη φορά τότε είχαμε υπονοήσει ότι θα ακολουθήσει το Q η ποσοτική χαλάρωση. Το Δεκέμβρη είχαμε πει 30% περίπου πληθωρισμός και ε, ανάπτυξη χαμηλή. Έκτοτε όμως έχουν προκύψει πάρα πολλά. Σας είπα ότι ε, η ανεργία είναι χαμηλότερη από το 2008 και πάνω από 11 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, ε, προέκυψαν σε λιγότερα από 6 χρόνια. Ε, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλές θέσεις εργασίας και νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην νομισματική πολιτική. Γιατί δεν υπήρχαν πολλές άλλες πολιτικές που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια Παράλληλα και συμφωνώ μαζί σας, ε, το ποσοστό πληθωρισμού λόγω παρεμβαλόμενων παραγόντων, λόγω γεωπολιτικής αστάθειας, αυτά οδήγησαν στο να μην έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Και έτσι σήμερα κάνουμε τα ίδια με την ίδια αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ε, φτάσουμε το στόχο μας ε, του πληθωρισμού. Ο κύριος Φερνάνδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους της ομάδας μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν ήμουν βουλευτή όταν εσεί ε, αναλάβατε, ενώ ο συνάδελφο Φέρμπερ ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα χρόνια είχαμε ε, πολύ καλή συνεργασία στα πλαίσια της ανεξαρτησίας βέβαια της ΕΚΤ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για την αναθεώρηση του πλαίσιου της νομισματικής πολιτικής. Το σημερινό πλαίσιο το έχουμε από το 2003. Από τότε μέχρι σήμερα, εσείς, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δράσατε σε αυτό το πλαίσιο αλλά επίσης ότι κάνατε και καινοτομίες στο δικό σας πλαίσιο δηλαδή. Μπορεί να μην αναθεωρήθηκε το ίδιο το πλαίσιο, παρόλα αυτά πήρατε και άλλα μέτρα. Έχετε μιλήσει πρόσφατα για τη συμμετρία του στόχου σταθερότητας τιμών. Μία συμμετρία η οποία με τον σημερινό ορισμό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν είναι ξεκάθαρη. Και γίνονται διάφορες ακαδημαϊκές συζητήσεις για την αναγκαιότητα ε, τη σταθερότητα των τιμών, όχι τόσο ε, με μέτρα πληθωριστικά, αλλά όσον αφορά τις τιμές αυτές καθε αν πρέπει να βάλουμε ενεργητικού, αν πρέπει να βάλουμε για τα κίνητα. Γνωρίζετε επίσης ότι γίνονται συζητήσεις και για τη δυνατότητα έκδοσης ε, digital currencies, δηλαδή να επιτρέψει η ΕΚΤ να έχουν ε, ε, λογαριασμούς ε, τέτοιους στις τραπεζές τους οι πολίτες, ώστε έτσι να διευρυνθεί κάπως το φάσμα των δυνατοτήτων. Η επόμενη πρόεδρος, δεν ξέρω κατά πόσο θα κοιτάξει να αναθεωρήσει το πλαίσιο. Πάντως θέλω να σας ρωτήσω όχι τόσο σε σχέση με το τι έγινε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά για το μέλλον. Εσείς πώς βλέπετε την νομισματική πολιτική στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Uh, Δύσκολη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπατε για τη συμμετρία. Η συμμετρία είναι πολύ σοβαρό στις αντιδράσεις που προβλέπουμε, διότι ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών ήταν ε, περίπου στο 2 και κάτω από το 2%. Αυτό δημιούργησε κάποιες παρανοήσεις ότι θα ήταν πιο δυναμική η αντίδρασή μας σε επίπεδα πληθωρισμού πάνω από το 2%. και ότι θα αντιδρούσαμε μετά σε ποσοστά κάτω του 2%. Υπήρχε λοιπόν φαίνεται διαφορετική ε, προσδοκία για το πώς θα αντιδράσουμε σε χαμηλό ή υψηλό πληθωρισμό. Όμως ως προς τη συμμετρία, αυτό που σημαίνει συμμετρία είναι ότι με την ίδια αποφασιστικότητα, πυγμή ε, και δυναμισμό θα αντιδράσουμε είτε είμαστε πάνω είτε κάτω από το στόχο του 2% που έχουμε. Αυτό σημαίνει συμμετρία. Δηλαδή ο πληθωρισμό μπορεί να πάει πάνω από το 2% ή κάτω από το 2%. Δεν είναι ο στόχο ε, του ορισμού των τιμών. Απλώ σημαίνει πώ θα αντιδράσουμε. Ω προ το πώ αντιδράμε εμεί είναι το θέμα. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να πούμε Πώ θα διαμορφωθεί η νομισματική πολιτική στο μέλλον. Νομίζω ήταν σαφέ από την εισαγωγική μου παρέμβαση ότι η νομισματική πολιτική έχει κάνει τη δουλειά τη, θα συνεχίσει να την κάνει. Όταν λέω ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να έχει ισχυρότερο ρόλο, δεν εννοώ καθόλου ότι η νομισματική πολιτική έχει εξαντλήσει το δυναμικό της είτε τα εργαλεία που διαθέτει την, την αποτελεσματικότητά της θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, αλλά αν οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι ενεργές, οι νομισματικές πολιτικές θα κάνουν τη δουλειά τους γρηγορότερα και με λιγότερες, παρα... Ε, παρενέργειες. Αυτό επιδιώκαμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκαρικάνο. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη, στην τελευταία σας παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω που το 2012 σώσατε το ευρώ όταν δεχόταν στιγμή επίθεση από το χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε. Στο Λάνκαστερ, στον Νίκο Λάνκαστερ, ήταν διάσημα τα λόγια σα από εκείνη την ομιλία. Όταν είπατε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για το κοινό νόμισμα και δεν απογοητεύσατε του Ευρωπαίου πολίτε. Σα ευχαριστώ λοιπόν και φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοί μου θα κάνουν το ίδιο. Ωστόσο θα κατανοείτε ότι σε κανέναν δεν αρέσει να έχει ένα νόμισμα που χρειάζεται διάσωση. Το είπατε και στην εισαγωγική ομιλία σας, στο δεύτερο εμισή. E είπατε ότι παραμένουν κάποιες αδυναμίες στην Ευρωζώνη. Για αυτό το δεύτερο μέρος της παρουσίασης, λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικού τριγμού και να χρειάζεται πάλι διάσωση το ευρώ και η ευρωζώνη. Αλλά τέσσερα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μα. Κάποια στιγμή τα εξετάζει η Επιτροπή, κάποια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί ποιε προτεραιότητε έχετε. Πρώτα απ' όλα το σχέδιο διάσωση και κάλυψη των εγγύσεων των καταθέσεων. Κάτι που απασχολεί την Επιτροπή μα. Μετά το SBBS, το ενιαίο σύστημα περιουσιακών του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα περάσει και από το Συμβούλιο. Μετά ο προπολογισμό της Ευρωζώνης, με την ενδεχόμενη εγγύηση για την ενέργεια των νέων. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε ένα ομοσπονδιακότερο, τέλος πάντων ευρωπαϊκότερο επίπεδο για όλα αυτά. Το είπε και η κυρία Φονταλάιν, τουλάχιστον επενήθηκε. Και μετά τι θα γίνει με τις κρατικές τράπεζες και τα χαρτοφυλάκια τους. Πώς θα γίνουν αυτά πιο ποικίλα ώστε να ε, μην ε, κινδυνεύουν. Ποιες είναι οι σχετικές σας προτάσεις. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα πρέπει να διασώσουμε ή όχι στο μέλλον και τι από αυτά βλέπετε ως το πλέον σημαντικό. Και επιπλέον πολλοί από εμά ανησυχούν για μια μεγάλη χώρα της Ευρωζώνης, την ξέρετε καλά, την Ιταλία. Εδώ και 30 χρόνια δεν έχει ανάπτυξη τι συμβαίνει με την Ιταλία, πόσο να ανησυχούμε, γιατί δεν αναπτύσσεται και τι θα έπρεπε να κάνει για να αναπτυχθεί. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα από, τους ε, από τις μεγαλύτερες απειλές για την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που θυμήσατε το 2012 έχει γίνει πρόοδο. Έχει γίνει πρόοδο στην οικοδόμηση τη νομισματικής και Οικονομική Ένωση. Ήταν πραγματικά επί τη ουσία η πρόοδο αυτή. Και είναι επίση σημαντικό όταν κανείς επιμένει στις σημερινές αδυναμίες να μην παραγνωρίζει τι σημαντική πρόοδο έχει, έχει ήδη επιτελεστεί. Θυμηθείτε ότι ακριβώ εκείνη τη χρονιά, τον Ιούνιο του 2012, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε την... να εξετάζει την πρόταση για την Τραπεζική Ένωση. Πολλά έχουν γίνει λοιπόν. Πολλά πρέπει να γίνουν και βραχυπρόθεσμα του ερχόμενου έξι μήνε και ένα χρόνο. Αλλά πρέπει απλώ να συμπληρωθούν τα κομμάτια αυτών που ήδη έχουν εγκριθεί. Δηλαδή να αποπερατωθεί η Τραπεζική Ένωση, το σύστημα εγγύηση των καταθέσεων και τα άλλα τμήματα τη Τραπεζική Ένωση. Κάποια πράγματα που έχουν ήδη εγκριθεί πρέπει να γίνουν κάπως λειτουργικότερα, κάπως πιο εύχρηστα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που λείπουν στο μηχανισμό διάσωσης, όπως η ρευστότητα σε συνδυασμό με τη διάσωση και κάποια άλλα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν είναι αυτά που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ε, εγκριθεί μάλλον. Μετά απομένει και η αποπεράτωση της, κεφαλόχη, της ε, Αγορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε ότι θα πρέπει το ευρώ να έχει έναν ισχυρότερο ρόλο στο διεθνές προσκήνιο, μοιάζει σαν να λέμε ότι θέλουμε απλώς να το προωθήσουμε, να το διαφημίσουμε. Το πρώτο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι η ένωση των κεφαλαιογορών. Γιατί το δολάριο έχει τέτοιο προεξάρχοντα ρόλο. Γιατί υπάρχει ένωση κεφαλαιογορών. Και είναι ένα σαφές ε, ε, όπλο ισχυρό και ασφαλέ όπλο. Βεβαίω το όλο πακέτο μέτρων είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο, θα χρειαστεί χρόνο. Όμω το πρώτο πράγμα, κατά πρώτον, είναι ήδη να ολοκληρώσουμε ότι έχει εγκριθεί ή σχεδιαστεί χαραχθεί. Α πούμε για την Ένωση των Κεφαλαίων χρειάζεται περισσότερη. Ε, ε περισσότερη ε, αρμονία στον ε, στην ομοθεσία των κατών μελών για τις περιπτώσεις αφαιρεγκαιότητα, τις διαδικασίες αφαιρεγκαιότητα και πτώχευσης. Έπειτα, πρέπει να είμαστε και φιλοδοξότεροι. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά αυτό που έχει σημασία εδώ και παρεμπιπτόντω αυτά δεν είναι μόνο σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά είναι σημαντικά για να τονώσουμε και την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, των ιδιωτών θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομική θέση και κατάσταση, το οικονομικό κλίμα της Ευρωζώνης. Τα άλλα σημεία που αναφέρατε, το μηχανισμό επανα... αντασφάλισης, τον ε, μηχανισμό εγγύσης των καταθέσεων, αυτά είναι θεμελιώδου σημασία για να αντιμετωπίσουμε τι αδυναμίε τη Νομισματική Ένωση. Δεν υπάρχει νομισματική ένωση στον κόσμο που να μην έχει δημοσιονομική πολιτική. Η πρόοδο λοιπόν που έχει επιτελεστεί ήδη είναι σημαντική. Η Ευρωζώνη και το ευρώ είναι πολύ ισχυρότερα. Η αποδοχή από το κοινό, από την κοινή γνώμη είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, υψηλότερη από ποτέ νομίζω, βάσει των δημοσκοπήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ερευνών, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και δεν είναι η πολιτική στόχη βραχυπρόθεσμη, είναι μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Γι' αυτό πρέπει η, η σαφής, από την αρχή να υπάρχει μια σαφής πολιτική δέσμευση. Η δεύτερη ερώτηση είναι ιδιαίτερα πολυδιάστατη. Αφορά πολλές διαφορετικές πτυχές. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι με μια απλή κουβέντα σε αυτή τη φάση. Και δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αλλά και μια σειρά από άλλες χώρες. Και έχει να κάνει με την ατζέντα των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Δεν καθορίζουν μόνο τον προπολογισμό. Οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και τομέων έχουν να κάνουν με μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ας πούμε. Πολύ σημαντικό, αλλά και για την αγορά των προϊόντων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτά είναι επίσης εξίσου σημαντικά, για να μην πω περισσότερο. Και κάποια άλλα που ίσως χρονικώς να πρέπει να προηγηθούν. Ο δικαστικός κλάδος, το εκπαιδευτικό σύστημα, το μέσο της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε χώρα εάν έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη, όπως και θα έπρεπε. Ευχαριστούμε. Ο Φιλίπ Λαμέο, από τους Πράσινους. Καλησπέρα σας. Ε, εγώ εξελέγηνα ως ευρωβουλευτής όταν αναλάβατε εσείς, άρα δηλαδή είχαμε τη χαρά αυτά τα τελευταία οκτώ χρόνια να τα περάσουμε μαζί. Ε, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπερασπιστήκατε αυτό το κοινό αγαθό, το ευρώ. Ε, και για ό,τι και αν είχε σχεδιαστεί, εξακολουθεί να υπάρχει το ευρώ. Αν εξαφανιζόταν το ευρώ θα ήταν μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ε, και εσείς κάνατε ό,τι μπορούσε. Κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για έλλειψη αποφασιστικότητα. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Ε, κατ' ουσίαν τι κάνατε. Την ε, κρίση την καλύψατε με ένα τσουνάμι και χρησιμοποίησατε την στάνταρ μέθοδο, δηλαδή κατ' ουσίαν, όπως σας είπα, πλημμυρίσατε με ρευστότητα το χρηματοπιστωτικό σύστημα εμείς ε, δεν συμφωνούμε μαζί σας ε, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Αν δούμε λιγάκι τις ανισότητες και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία το οικολογικό αποτύπωμα και την κλιματική κρίση, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο στο τομέας ήταν αποτελεσματικός ε, διανομέας κονδυλίων. Μετά την κρίση δεν βλέπουμε να έγινε αποδεκτό το μάθημα. Μία άλλη μέθοδος ε, είναι τα χρήματα που μεταφέρονται ξαφνικά με αεροπλάνα, με ελικόπτερα, ε, είπατε ότι διερωτηθήκατε κατά πόσον αυτό πράγματι θα ήταν μια σωστή νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική. Τελικά όμως καταλήξατε σε αυτήν. Πάντως, ε, βλέποντας λιγάκι τις ε, πολιτικές τις οποίες εφαρμόσατε, αυτή την πολιτική που μεταφέρονται, των χρημάτων που μεταφέρονται με αεροπλάνα, αυτή είναι η πολιτική των πλουσίων. Το αντίθετο βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν δεν γίνει όμως αυτό θα προέκυπτε μια χειρότερη κατάσταση και αυτή θα επιτείνει την ανισότητα. Αν όμως οι ε, δύο λύσεις είναι QE, e, quantitative easing, ποσοτική χαλάρωση ή το να μην κάνει κανείς τίποτα, αυτό δεν είναι ένα σωστό δίπολο. Εγώ ε, θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας. Το ένα στοιχείο είναι η ανισότητα και το δεύτερο στοιχείο είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και το κλιματικό αποτύπωμα. Είπατε ότι δεν είμαι εγώ εκείνο που θα αποφασίσει, αλλά το θέμα είναι ότι η ρευστότητα έχει μεταφερθεί σε περιοχές όπου ήταν επιζήμιο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις ανισότητες, πολύ σωστά υπενθυμίσατε και το έχουμε συστήσει αυτό επανειλημμένα, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η ποσοτική χαλάρωση ε, βελτιώθηκε γιατί η ανεργία μειώθηκε και αυτό είναι μια βασική πηγή ανισοτήτων. Είναι σαφές ότι όταν ε, αυξάνονται οι τιμές, ε, αυτοί που αποφελούνται είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα. Υπάρχει βέβαια και ένας μηχανισμός ε, αναδιανομής, αλλά αυξήθηκαν πράγματι και οι τιμές ε, των ε, σπιτιών, της στέγασης. Όμως ε, το να δημιουργηθούν όλες αυτές οι θέσεις απασχόλησης, σας λέω, αυτό σήμαινε μείωση των ανισοτήτων. Η ανεργία είναι εκείνη που προκαλεί τις ανισότητες. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, αυτά δεν ισχύουν μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά και για όλες τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Δηλαδή, εφαρμόζει κανείς νομισματική πολιτική, χορηγώντας ρευστότητα μέσα από τα κανάλια που υπάρχουν. Στην Ευρώπη, Ευρώπη έχουμε τις τράπεζες που κυριαρχούν. Άρα, αν θέλετε, είναι μια οικονομία που βασίζεται στις τράπεζες και η δική μας η νομισματική πολιτική ε, λειτουργεί μέσα από το κανάλι του δανεισμού στις τράπεζες. Ε, στις ΗΠΑ το σύστημα λειτουργεί περισσότερο με τις αγορές. Αυτά τα δύο συστήματα υπάρχουν. Όπως είπατε, είναι άραγε αυτός ο καλύτερος τρόπος για να χορηγεί κανείς ρευστότητα αν έχει κατά νου στόχους όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή η μείωση των ανισοτήτων με αποτελεσματικότερο τρόπο. Ίσως όχι, ίσως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι και πράγματι ορισμένες από τις νέες απόψεις που έχουν προκύψει για την αφισματική πολιτική όπως το MMT ή το τελευταίο έγγραφο ε, που παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων με τον καθηγητή κύριο Φίσερ και από άλλου, προτείνουν διαφορετικού και διάφορου τρόπου για να χορηγούνται χρήματα στην οικονομία. Αυτά ε, είναι προφανώ ε, νέε απόψει. δεν έχουν συζητηθεί ακόμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, Ω εκ τούτου θα πρέπει να τι εξετάσουμε αυτέ τι απόψει, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί. Και όταν, αν τις δει κανεί έτσι λίγο πιο προσεκτικά αυτέ τι απόψει, θα διαπιστώσει ότι αυτό το καθήκον του να αναδιανέμονται δαπανώνται χρήματα, αυτό κατ' ουσίαν είναι δημοσιονομικό καθήκον. Δηλαδή, τι είναι, είναι απόφαση τράπεζα, όχι και, ε, απόφαση κυβέρνηση με συγχωρείτε, και όχι κεντρική τράπεζα. Εσείς λέτε η κεντρική τράπεζα πρέπει να αποφασίζει ποιο θα λαμβάνει τα χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με αυτέ τι νέε απόψει, αλλά ένα βασικό θέμα είναι η πολιτική διακυβέρνηση σε σχέση με αυτέ τι νέε απόψει. Αυτό πρέπει να δούμε ο Αντώνιο Ρινάλντι από το ε, κόμμα, από την ε, ομάδα ID. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ιταλικά. Πρόεδρε Ντράγκη, είμαι πεπισμένο ότι κάποια μέρα η ιστορία θα σα αναφέρει ω τον, τον άνθρωπο που έσωσε το ευρώ. Εάν εσεί από την αρχή δεν είχατε αναλάβει έκτακτα μέτρα και την έκτακτη απόφαση της ε, ποσοτικής χαλάρωσης και της τόνωσης του νομίσματος, θα ήμασταν σήμερα σε συνθήκες πολύ χειρότερες. Πραγματικά λοιπόν σας αξίζει παράσημο ε, για τη διάσωση αυτή. Παρ' όλα αυτά ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια και προσωπικά. Έχετε στην κεντρική τράπεζα κάποιες γραπτές αρμοδιότητες που προκύπτουν από το ίδιο το καταστατικό της τράπεζας, όπως έχει καταρτιστεί. Και θα έλεγα ότι έχετε καταφέρει και κάποια. Δεν μπορείτε να κάνετε μάλλον και θαύματα. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξή. Πότε νομίζετε ότι μπορεί μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπω η Ευρωπαϊκή να εξακολουθεί χωρίς τις ανάλογες δημοσιονομικές πολιτικές από το κάθε κράτος μέλος πώς μπορεί να συνεχίσει να τα καταφέρνει και να τα πηγαίνει καλά. Ε, γιατί όλη η οικοδόμηση της Ευρωζώνης πρέπει να αλλάξει τελείω. Και μια ερώτηση λίγο σπρόκληση, Πρόεδρε. Στην 1η ε, Νοεμβρίου, την επόμενη μέρα, the day after όπως τα λέγαμε, μπορείτε να μας πείτε Ποια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να έχουμε για να καταφέρουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε μια ευρωζώνη που δεν θα έλεγα να είναι η τελειότερη ή η άριστη, αλλά να είναι κοντά στο ιδανικό που θέλαμε να πετύχουμε. Διότι ξέρουμε ότι έχουμε άλλες κεντρικές τράπεζες που είναι διαφορετικά διαθρωμένες. Δεν είναι οι τελευταίοι δανειστές μόνο, είναι και άλλοι στόχοι τους, ξέρω εγώ, να ελέγχουν τον πληθωρισμό ή το ποσοστό της απασχόλησης. Σε πολλά συντάγματα άλλωστε ε, προβλέπεται αυτό ως ε, θεμέλιο και ως στόχος. Αλλά Πώς μπορεί το ευρώ να γίνει ξαφνικά ε, αυτός που θα διασώζει μέσα σε ένα πλαίσιο που τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και σωστά διαρθρωμένα. Την 1η Νοεμβρίου λοιπόν, την επόμενη μέρα, μπορείτε να μας πείτε πώς θα θέλατε να μοιάζει η Κεντρική Τράπεζα για να κάνει τη δουλειά της. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω στα Ιταλικά, αλλά μάλλον θα προτιμήσω τα Αγγλικά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τους επένους σας και τα καλά σας λόγια, αλλά να πω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει μετά την 1η Νοεμβρίου. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ του να έχουμε ένα ισχυρό όπλο για τη δημοσιονομική, ως, ε, τη δημοσιονομική πολιτική, μάλλον ω ισχυρό όπλο. Ή καλύτερα να υπάρχει δημοσιονομικό συντονισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι οι δημοσιονομικοί κανόνε σε επίπεδο κάθε χώρα θα πρέπει να μην είναι τόσο ε, προκυκλικοί, να ασχολούνται με τους οικονομικούς κύκλους δηλαδή μόνο. Ε, η εμπειρία που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποδείξει ότι ε, ήταν αφοσιωμένα και σχεδιασμένα με βάση τους οικονομικούς κύκλους. Σε καιρούς προκρίσης, πολλές χώρες είχαν ε, ασχοληθεί με το έλλειμμά τους κυρίως, το είχαν αυξήσει πάρα πολύ, χωρίς μαξιλαράκια, χωρίς προστατευτικά. Ε, και όταν έφτασε η κρίση, κάποιες χώρες που είχαν αυτά τα μαξιλαράκια τα χρησιμοποίησαν και μπόρεσε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, κυρίως ε, σώζοντας τις τράπεζες τους. Μην ξεχάσουμε ότι σε κάποιες χώρες οι τράπεζες πραγματικά ε, κατέρευσαν στο πρώτο μέρος της κρίσης το 2010, 9 Και τις βοήθησαν πάρα πολλοί οι κυβερνήσεις με τις αγορές τους και τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Γιατί υπήρχαν τα μαξιλαράκια. Σε χώρες χωρίς μαξιλαράκια δεν διασώθηκαν οι τράπεζες. Οπότε ξεκίνησε μια κρίση χωρίς τέλος, η οποία συνεχίζεται και είναι υποκείμενη τρόπον την άμεση σήμερα. Πολλά από τα μαξιλαράκια, λοιπόν, σε πολλές χώρες επέτρεψαν στην ε, δημοσιονομική πολιτική να προσαρμοστεί αναλόγως, ακριβώς επειδή υπήρχαν ε, τα μέτρα προφύλαξης. Όμω, είναι αρμοδιότητα δική σα περισσότερο του Ευρωκοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα κάνετε αυτά. Δεν μπορούμε να τα αποφασίσουμε εμεί ω Κεντρική Τράπεζα. Το δεύτερο που ρωτήσατε για τη δημιουργία ενό δημοσιονομικού εργαλείου που ως βασικό στόχο θα πρέπει να έχει την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Αυτό είναι ένα μακρόπνο εγχείρημα και είναι και πολιτική πρόκληση. Γι' αυτό δεν είναι και σαφές ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε τώρα μια πολιτική δέσμευση από κάποια πλευρά. Για να λειτουργήσει όμως τέτοιο ένα εργαλείο θα πρέπει να έχει στόχο τη σταθεροποίηση, να έχει και τον κατάλληλο όγκο, μέγεθος, αλλιώς δεν θα είναι αξιόπιστο και να είναι και σχεδόν αυτόματη λειτουργία του, να χρησιμοποιείται αμέσως, ε, Γι' αυτό και ο αυτόματος χαρακτήρας στη χρήση του είναι σημαντικός. Παραδείγματα από άλλες νομισματικές ενώσεις θα μπορούσαν να είναι και πολύ χρήσιμα Κάτι ανάλογο μάλλον συμβαίνει και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτήν την δημοσιονομική, ε, επανα, τον οικονομικό, δημοσιονομικό επανασχεδιασμό χρειαζόμαστε για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τώρα για την εντολή μας, τις αρμοδιότητές μας. Δεν θα ήταν καλύτερα λέτε να είχαμε διπλή εντολή αντί μόνο τη σταθεροποίηση των τιμών. Η ερώτηση αυτή έχει τεθεί και απαντηθεί επανειλημμένως. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για να ε, σχεδιάζουμε τη δική μα την εντολή. Δεν τι αποφασίζουμε εμεί. Εσεί οι νομοθέτε τι αποφασίζετε. Αλλά από πρακτική σκοπιά έχουν γίνει και κάποιε έρευνε τα προηγούμενα χρόνια που δείχνουν. Δεν ξέρω πόσο επίκαιρε είναι οι έρευνε αυτέ, αλλά δείχνουν ότι αν δει κανεί τα πράγματα εκ των υστέρων, το αν έχει κανείς μία ή δύο εντολές, στο κάτω-κάτω της γραφής, το ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει. Δεν είναι και τεράστια η διαφορά. Διότι αν δείτε πώ αντιδράσαμε βάσει αυτή τη λειτουργία, αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν πλήρη απασχόληση στην Ευρωζώνη. Ακόμη και αν έχουμε πετύχει κατά το ίμιση του στόχου τη σταθεροποίηση των τιμών. Δηλαδή, δημιουργήσαμε συνθήκε τέτοιε ώστε να υπάρχει σταθερότητα στι τιμέ στο μέλλον και έχουμε τουλάχιστον ονομαστικό ποσοστό ε, για την απασχόληση που φτάνει επίπεδο του παρελθόντο. Πολύ καλά. Ακόμη δεν έχουμε δει τη σταθερότητα των τιμών που θέλαμε, αλλά θα γίνει και αυτό μελλοντικά από ό,τι φαίνεται. Πάνε δηλαδή παράλληλα με διαφορετικό ρυθμό. Δεν είναι σαφέ όμω να διακρίνουμε το τι θα είχαμε πετύχει αν είχαμε διπλή εντολή αντί για τη μία που έχουμε τώρα και για, τα ποσοστά, για τι ισοτιμίε τώρα. είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Ε, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία, όλες οι κεντρικές τράπεζες λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, μάλλον, μας ε, δεσμεύει η, η ε, απόφαση του G20, οπότε εκεί υποχρεούμεθα να σεβαστούμε τις αποφάσεις του G20. Δεν νομίζω ότι το ευρώ είναι πιο αδύναμο σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου ως προς την πτυχή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φανόφερφελτ, από το ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Ντράγκη, εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ και σας εύχομαι ήδη από τώρα ό,τι καλύτερο για την περίοδο μετά την ε, εντολή σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να κάνω τρεις δηλώσεις και μετά τα σχόλιά σας παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα για τις ισοτιμίες με τις αποφάσεις του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, δύσκολα μπορώ να φανταστώ αυτά τα μέτρα να έχουν πραγματικά μεγάλες επιπτώσεις στις επενδύσεις και στην κατανάλωση από πλευράς των καταναλωτών. Και ανησυχώ για αυτά που είπατε για την οικονομική ανάπτυξη. Οπότε υποθέτω ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι που έχουν να κάνουν με τις ισοτιμίες, προλαμβάνοντας ίσως ε, το γεγονός ότι και άλλες κεντρικές τράπεζες ε, θα πάνε ε, προς το δρόμο της ποσοτικής χαλάρωσης και εσείς αντιδράτε εκ των προτέρων για να προκαταλάβετε αυτές τις δράσεις. Δεύτερον, αρχίζετε επαναγορά πάλι, είπατε 20 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα και λέτε επίσης ότι μπορεί να πάτε και ακόμα παραπέρα. Δηλαδή μπορεί η ΕΚΤ να αγοράσει πιο επικίνδυνες ε, μετοχές, ιδιωτικά κεφάλαια. Και τρίτον, αναφερθήκατε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την συμφωνία που έχετε εκεί όσον αφορά το ρόλο της δημοσιονομικής ε, πολιτικής, που θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Μάθαμε για την ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες και είδαμε ότι υπήρξε διαφοροποίηση στην ψηφοφορία. Τι έχετε να πείτε και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα. Αν είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές μας, ρωτάτε. Λοιπόν, τι να σας πω. Κοιτάξτε μόνο πόσες θέσεις απασχόλησης έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Ή δείτε, είναι διάφορα τέτοια στοιχεία, ανεργία κτλ. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα από το 2014 και αυτά που αποφασίστηκαν τον Ιούνιο του 2019, όχι τα τελευταία δηλαδή, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό και στις δύο περιπτώσεις είναι 2,2% συσσωρευτικά από το 2016 μέχρι το 2021. Άρα είμαστε σίγουροι ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα μας. Δεύτερον, όταν οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ μείωσαν τις προοπτικές, πριν από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, αυτό οδήγησε στις αποφάσεις μας και οι προβολές αυτές ε, βασίζονται σε ένα σύνολο επιτοκίων που ήδη αντικατόπτριζαν ε, κάποιες προσδοκίες για δράση της ΕΚΤ δεδομένων ε, των ε, κακών ε, προβλέψεων. Αν δεν είχαμε δράσει, θα έπρεπε να είχαμε μειώσει ακόμα περισσότερο τα επιτόκια και τις προοπτικές μας για την ανάπτυξη. Και αυτό θα ήταν ένας φαύλος κύκλος που θα μας απομάκρυνε τελικά από την εντολή μας. Τώρα το τρίτο που ρωτήσατε για τις συζητήσεις. Μα υπήρξε σαφής πλειοψηφία υπέρ της δέσμης μέτρων που υιοθετήθηκαν τελικά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Χωσέ από την ΚΟΕ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Πορτογαλικά, αν δεν σας πειράζει. Δύο σχόλια και δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή νομίζω όλοι συμφωνούν για το ρόλο που έχει η νομασματική πολιτική στο να αποφύγουμε την κατάρρευση της Ευρωζώνης. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την εντολή της συμπεριφέρθηκε όπως άλλες κεντρικές τράπεζες με διαφορετικές εντολές. Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό για σας προσωπικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά όχι σε σχέση με την αντίδραση της τράπεζας ε, στις αρχές της κρίσης. Ή σε, αντίδραση, σε αντιδιαστολή με το τι συνέβη στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τη ΦΕΤ. Πάντως, είναι σημαντικό να μιλάμε για δημοσιονομικά εργαλεία αντικυκλικά, κάτι που φάνηκε ότι χρειαζόταν στην Ευρωζώνη μετά την ε, κρίση. Αυτό ήταν θετικό, αλλά δεν μπορούμε να περιορίζουμε τη συζήτηση σε χώρε με μικρότερο περιθώριο λιγμών ε, στη δημοσιονομική πολιτική. Λόγω χάρη η χώρα από την οποία προέρχομαι μείωσε το επίπεδο του ΑΕΠ κατά κάποιε ποσοστιαίε μονάδε και αυτό το έκανε με την θετική διαχείριση κάποιων κρατικών λογαριασμών βεβαίω Άρα η μακροοικονομική πολιτική δεν αρκεί μόνο. Χρειάζονται και πολιτικές ισότητας, περιβαλλοντικές πολιτικές, πολιτικές ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν διαθετικά προβλήματα. Άρα ήθελα να μου πείτε τι θεωρείτε ότι οι υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης πρέπει να κάνουν. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούν και το, το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων για να καταρτήσουν αντικυκλικά δημοσιονομικά εργαλεία. Και έπειτα επειδή υπήρξαν αντιφατικά σχόλια εδώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το θέμα αυτό, ήθελα να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι πρόσφατε εξελίξει στις αγορέ εργασία και οι συστάσεις που έγιναν από τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση της ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας με ε, περιορισμό των συλλογικών συμβάσεων στην αγορά εργασίας και των σχετικών ε, διάβλων τους. Δεν είναι κάτι που δυσχεραίνει τα πράγματα και κάνει τελικά μικρότερη πιθανότητα να αυξηθούν κάπως οι μισθοί και να υπάρχει ε, χειρότερη υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής εν τέλει. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Είναι αρκετά σαφές ότι χώρες με ψηλό χρέος θα πρέπει να είναι συνετές στη δημοσιονομική τους πολιτική για να μην επέλθει από σταθεροποίηση. Αστάθεια στη συνολική ισορροπία γιατί σήμερα τουλάχιστον έχουν πρόσβαση στι χρηματαγορέ. Εάν δούμε τι γινόταν πριν από λίγα χρόνια, δεν ήταν καλό αυτό για την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι' αυτό είπα ότι οι δημοσιονομικοί κανόνε πρέπει να αναθεωρηθούν. Οι δημοσιονομικοί κανόνε που είχαμε ω τώρα ήταν αποτελεσματικοί, ήταν και λογικοί για αρκετά χρόνια. Τώρα όμως λογική ακόμα είναι, αποφεύγουν την υπερβολική σώρευση χρέου, όμω δεν είναι πλέον το ίδιο αποτελεσματική, δεν είναι προσαρμοσμένη στι ανάγκε αντιμετώπιση των ε, κυκλικών επιπτώσεων τη οικονομία. Εκεί χρειάζεται η αναθεώρηση. Όμω γι' αυτό ακριβώ και για χώρε με σωστή δημοσιονομική πολιτική, συνετή, ένα κεντρικό εργαλείο ε, σταθεροποίηση δημοσιονομική είναι τόσο σημαντικό. Υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν ασυμμετρικά σοκ. Εκεί πρέπει να έχουν τα κατάλληλα μαξιλεράκια, τις κατάλληλες προφυλάξεις. Και υπάρχουν και άλλοι τριγμοί, άλλοι κλειδονισμοί που ασταθεροποιούν συνολικά την Ευρωζώνη. Εκεί τα κεντρικά δημοσιονομικά εργαλεία θα μπορούσαν να είναι σημαντικά. Ταυτόχρονα, τίνουμε να το παραγνωρίζουμε, διότι έχει γίνει πολύ πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις είναι το μόνο εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οικονομίες για να σχεδιάσουν και να στοχεύσουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Δεν αναφέρομαι ειδικό στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Μιλάω για την ανταγωνιστικότητα, μιλάω για την ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, του εκπαιδευτικού συστήματος, Εκεί όλος ιδιαίτερε χώρε που έχουν ένα σύστημα και μια διαδικασία ανάπτυξη πιο ευάλωτη, πιο εύθραυστη, πρέπει να δουν και αυτές τις μεταρρυθμίσει. Τώρα για την ερώτησή σας, για το κατά πόσον υπήρξε τέτοια πρόταση διάλυσης, δεν, δεν το γνωρίζω. Τι είναι αυτό? Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα ο δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε λίγο στον πρώτο και δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Θα θυμίσω ότι έχουμε όριο. Τέσσερα λεπτά για την ερώτηση, το σλότ, και τρία λεπτά για την απάντηση. Ιδάλλως δεν θα προλάβουμε. Λυπούμε. Ο κύριος Νίντερμαϊερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως και οι άλλοι και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντράγκη για την εξαιρετική δουλειά του. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από όλα αυτά που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Τρία θέματα να θίξω από την ομιλία σας. Το πρώτο είναι ότι άκουσα πολύ προσεκτικά τη νέα ανακοίνωση για την Forward Guidance και είναι νομίζω πολύ κοντά στην ανακοίνωση για τον πληθωρισμό. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναφέρεται ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο για νομισματική πολιτική αν χρειαστεί ότι μπορούμε να μετακινηθούμε προς τον α ή β δρόμο. Ε, ο, το περιθώριο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ε, πιστεύω ότι εννοείται δηλαδή ότι θα μπορούσαν να πράξουν και άλλα πιο αρνητικά επιτόκια. Και εάν ναι, ε, τότε ε, σε ποιο βαθμό η ρευστότητα θα μπορούσε να είναι ένα εμπόδιο στην πολιτική των αρνητικών επιτοκίων. Και κάτι τελευταίο. Με έχω εντυπωσιαστεί από το ότι συμπίπτει η ένταση στην αγορά εργασία, η ψηλή απασχόληση, ε, χαμηλός πληθωρισμός ε, και η, φέρποσα, η αυξημένες τιμές και υφέρπων πληθωρισμός σε ορισμένες χώρες βλέπουμε ότι δεν ισχύουν όμως ε, τα ίδια. Έχουμε υψηλές ε, τιμές στέγασης, ε, υψηλές τιμές στον χρηματοψηφιακό τομέα. Πώς ακριβώς εξηγείται αυτό. Ναι, η πρώτη ερώτηση είναι σαφώς ναι. Ε, έχουμε το στόχο του πληθωρισμού και κατά κάποιον τρόπο αυτός ανέκαθεν ήταν ο στόχος μας. Ο αυτό που κάναμε ήταν ε, ε, να διευκρινίσουμε την συμμετρία στις αντιδράσεις ε, και να μετακινηθούμε από καθοδήγηση όπου θα λέμε ότι ε, θα παραμείνουν οι τιμές σε αυτό το επίπεδο μέχρι την τάδε χρονική στιγμή, να κατευθύνουμε τα επιτόκια και να πούμε θα παραμείνουν τα επιτόκια σε αυτό το επίπεδο μέχρι να δούμε ότι ο πληθωρισμός συγκλίνει προς το στόχο μας. Όσον αφορά τώρα στη δεύτερη ερώτηση, αυτή αφορά να το πω αλλιώ. Ε, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στη ρευστότητα και τα αρνητικά επιτόκια. Δεν το βλέπουμε αυτό μέχρι τώρα. Επίσης, ε, η εισαγωγή του συστήματος δύο των βαθμίδων ε, θα έπρεπε να δώσει δυνατότητα της προϋποθέσεις όπου τα αρνητικά επιτόκια, η ανάγκη να περάσουν τα αρνητικά επιτόκια στους πελάτες θα είναι λιγότερο επίγουσα ε, σε σχέση με τη δυνατότητα της τράπεζας χορήγησης δανείων. Και το τρίτο θέμα είναι το pass-through. Είναι αλήθεια ότι η ονομαστική ανάπτυξη πραγματικά είναι πάνω από τους ιστορικούς ε, μέσους όρους σε όλες τις χώρες και κατά και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που έχει σχέση με την τρέχουσα κατάσταση είναι ότι ο δείκτης διάχυσης ε, στην ε, ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης είναι πολύ χαμηλός. Εδώ και αρκετό καιρό. Ως εκ τούτου εξακολουθούμε να μην βλέπουμε το να περνάμε από τις υψηλές ε, τιμές ε, των μισθών, σε υψηλότερες ε, τιμές ε, των αγαθών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την ζήτηση αν δούμε λιγάκι και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαπιστώσουμε εκεί ότι η κατανάλωση τα πάει πάρα πολύ καλά, λόγω του ότι και η απασχόληση τα πάει πολύ καλά. Η αγορά εργασίας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε το ίδιο να γίνει και στην Ευρωζώνη, όπου έχουμε δει ότι η αγορά εργασία ε, χάνει το δυναμισμό, βελτιώνεται στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά χάνει το δυναμισμό τη. Και σε ορισμένε ε, χώρε δεν βελτιώνεται η ανεργία, του αντίον το αντίθετο συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό το θέμα πρέπει να το προσέξουμε. Για την τελική ανάλυση το βασικό στοιχείο τη ανάκαμψη είναι η κατανάλωση. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπεντράκη, μάλλον θα χρειαστείτε τα ακουστικά. Πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε την οικονομική κρίση, αλλά και η σύνεση που διέσωσε το ευρώ, είναι ο κύριος λόγος που θα σας θυμούνται οι επόμενες γενιές και πιστεύω επίσης ότι αυτό εξηγεί και κάποιες από τις επιθέσεις προς το πρόσωπό σας, επειδή διασώζοντας το ευρώ έχετε διασώσει ουσιαστικά και το ευρωπαϊκό project. Μετά από αυτά τα καλά λόγια όμως θα πω κάποια που δεν είναι τόσο καλά. Το 2014 ανέλαβα ευρωβουλευτής. Η πρώτη ερώτηση που σας έθεσα ήταν πότε θα ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση με την εγγύηση των καταθέσεων. Ξέρω ότι η απάντησή σας ήταν περίπου ότι πρέπει να, πάρουν, να προχωρήσουν οι πολιτικοί σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από τον Μάριο Ντράγκη, με την αποφασιστικότητα και τη σύνεσή του, να δώσει το στίγμα σήμερα, πέραν από τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν. Πέραν. Και επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα. Σημερίζεστε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχετε θίξει ήδη συμμερίζεστε την άποψη που εκφράζεται και από κεντρικούς κυβερνήτες ε, τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχει αδυνατήσει εμπειρικά ο δεσμός ανάμεσα στο employment και στην αύξηση των μισθών. Και πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Μήπως είναι αποτέλεσμα των φοβερά αδύνατων εργατικών συνδικάτων λόγω της οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ και πάλι. Thank you. Um, σας ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και εδώ τώρα όχι μόνο η ΕΚΤ, αλλά και η Επιτροπή με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έδωσε μεγάλη όθηση στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης μέσω από τη δημιουργία του SSM. Αν πιστεύετε ότι ο υποπτικός ε, αυτός οργανισμός που υποπτεύει το τραπεζικό σύστημα ε, δημιουργήθηκε τόσο γρήγορα, ε, είναι σπουδαίο και κατάφερε να βοηθήσει από το μηδέν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εργάζεται με όλα τα ευρωπαϊκά υποπτικά συστήματα είναι μια τεράστια συνεισφορά στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Αλλά σίγουρα μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Για να έχουμε μια πραγματική Τραπεζική Ένωση πρέπει να μειώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών, κάτι το οποίο καθιστά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση ευάλωτη. Αλλά αυτό είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρο τη ολοκλήρωση ε, τη ε, Τραπεζική Ένωση είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Όσον αφορά πάντω την ΕΚΤ, εμείς θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ε, εποπτική λειτουργία. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τη σχέση της ανεργίας και του πληθωρισμού ενέργεια πληθωρισμός. Η σχέση σίγουρα έχει τροποποιηθεί τα τελευταία 15 χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε. Οι προοπτικές πληθωρισμού, οι ε, τιμές, η παγκοσμιοποίηση, η πίεση που ασκεί στο επίπεδο τιμών η παγκοσμιοποίηση κλπ. Η σχέση όμως παραμένει η σύνδεση. Εμείς, ενώ η ΕΚΤ, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ στηρίζουμε την έννοια αυτή η οποία βασίζεται στις εμπειρικές έρευνες. Και είναι κάτι που αποτελεί και την βάση της εμπιστοσύνης μας ότι τελικά ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον στόχο μας. Είναι η πεποίθησή μας. Ευχαριστούμε. Ε, Στεφανή Γιουγκορτόρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα καταφέρατε κατά τη διάρκεια της εντολής σας. Ε, πρόσφατα είπατε ότι συνολικά οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτιμούν τα θετικά από την οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίσατε ότι το 75% των κατοίκων της Ευρωζώνης είναι υπέρ του ευρώ και της νομισματικής ένωσης. Όμως η κοινή γνώμη είναι πολύ πιο επιφυλακτική όσον αφορά τη δομή και πρώτα απ' όλα το νομισματικό μηχανισμό που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που φαίνεται να βρίσκεται πολύ μακριά. Ε, κάτι ακατανόητο για τους ε, πολίτες και τις επιχειρήσεις. Εσείς λοιπόν πώς θα έρθετε πιο κοντά ε, στην κοινή γνώμη. Πώς δηλαδή η κοινή γνώμη, οι πολίτες θα καταλάβουν καλύτερα την πολιτική της ΕΚΤΕ. Πώς και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να σας ε, βοηθήσουμε περισσότερο σε, αυτό το, σε αυτή τη λειτουργία διαπαιδαγώγησης. Δεύτερον, είναι η ώρα του απολογισμού, κύριε Ντράγκη. Μετά από 8 χρόνια στην Προεδρία της ΕΚΤ, γιατί μπορείτε να πείτε ότι είσαστε περισσότερο περήφανος και γιατί είσαστε λιγότερο ικανοποιημένος. Τι είναι αυτό που σας κάνει πιο πολύ περήφανο και τι είναι αυτό που σας δυσαρεστεί περισσότερο από τη θητεία σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση πρώτα. Το ευρώ είναι αυτό που ε, συμβολίζει καλύτερα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί είναι αυτό που χρησιμοποιούν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορα εκλεγμένοι εκπρόσωποι εδώ και σε άλλα κοινοβούλια έχουν αναγνωρίσει ε, ότι έχουμε ευημερία, ε, κάτι το οποίο αποτελεί μία πρόκληση την οποία μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαι περισσότερο ισχυρή μαζί. Έχουμε φτάσει ε, σε ένα σημείο που δεν φανταζόμασταν όταν σχεδιάστηκε το ευρώ από 13% του ΑΕΠ ή του 92 εξαγωγές μας έχουν φτάσει στο 20%. Αλλά κυρίως οι αλυσίδες αξιών βρίσκονται παντού, όπως βλέπουμε. Και το βλέπουμε αυτό, ότι όταν μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση, αυτό είναι κάτι το οποίο μετακυλά και σε άλλες χώρες. Δεύτερον, το ευρώ αν δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, έχει βοηθήσει στη σταθερότητα τιμών. Και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Το θέμα της επικοινωνία στο οποίο αναφερθήκατε, έχει δύο διαστάσει. Η μία είναι ότι η επικοινωνία της ΕΚΤ στις διάφορες χώρες βασίζεται στη επικοινωνεί και στην βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Όπου μα στηρίζουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, η κοινή γνώμη είναι πολύ θετική απέναντί μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και να το διατηρήσουμε. Βέβαια υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση που λέει ότι δεν πρέπει κανείς να μιλάει μόνο με τις αγορές και με τις τράπεζες, αλλά πρέπει να μιλάει με τη γλώσσα του κόσμου. Και θα συμφωνούσα, αλλά εδώ θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί συγχρόνως. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι σε θέση να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας και της πολιτικής. Γιατί είναι πολύ εύκολο για να χρησιμοποιήσει κανείς τη γλώσσα του κόσμου τελικά ε, να μπει κανείς μέσα σε έναν κόσμο που δεν είναι αυτός της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά της πολιτικής. Και αυτό θα ήταν σε βάρος της αναξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε, ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κογκιόνι. Ελκ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Πρέπει να ξέρετε ότι οι πολιτικές σας ε, τον καιρό της κρίσης επενέθηκαν όχι μόνο από την Ευρωζώνη αλλά και εκτός Ευρωζώνης. Εγώ εκπροσωπώ μια χώρα εκτός της Ουγγαρίας και θυμάστε ότι η χώρα μου διασώθηκε ε, εγκαίρως ε, αλλά Επίσης για δεύτερη διαδικτική χρονιά ε, αναπτυσσόμεθα ε, γρηγορότερα από όλη την ε, Ένωση προς στιγμή. Μιλήσατε λοιπόν για αποτελεσματικές διαδικτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές πολιτικές και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και ήταν ένα σαφές δίδαγμα από την κρίση. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την κατάσταση των εκτός ευρωζώνης χωρών με διαφορετικές πολιτικές. Αποφασίσαμε πρώτα να συγκλίνουμε, να γίνουμε αρκετά δυνατοί και να έχουμε ένα ανθεκτικό σύστημα και να μπούμε στην Ευρωζώνη λίγο αργότερα ίσως, μεν, αλλά να αποφεληθούμε από τα διδάγματα του παρελθόντος. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά διδάγματα. Πώς εκτιμάτε στην την κατάσταση λοιπόν των χωρών αυτών και τι θεωρείτε για τις συνθήκες εισόδου στην Ευρωζώνη τις προϋποθέσεις μάλλον εισόδου. Διότι νομίζω ότι υπάρχουν νέες προϋποθέσεις και με την Τραπεζική Ένωση να έρχεται προς αποπεράτωση, αλλά δεν βλέπω να αλλάζουν σύντομα οι αιτήσει αυτές απαιτήσει. Όταν θα είμαστε αρκετά ισχυροί θέλουμε και εμείς να μπούμε στην Ευρωζώνη, αλλά την κατάλληλη ε, χρονική στιγμή. Ναι, αυτό που βλέπουμε να διαμορφώνεται μπροστά μας, η είσοδος στην Ευρωζώνη, στο ευρώ, περνάει από τρία κύματα. Πρώτα απ' όλα να είναι κανείς μέλος του RM2. Συνειδητοποιείται ότι σήμερα ότι μια χώρα μπαίνει όχι μόνο σε μια νομισματική ένωση, αλλά στις απαρχές μιας τραπεζικής. Και ενώ το πρώτο είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ταυτόχρονα, το άλλο έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την ε, ε, κεντρική με την ΕΚ την ίδια. Ε, το τι θα γίνει τώρα με μια χώρα που μπορεί να κάνει αίτηση για να, μπει, ε, να ξεκινήσει μάλλον μια, με μια συμφωνία στενής συνεργασία για την συμφωνία αυτή πρέπει να προηγηθεί μια διεξοδική αξιολόγηση από την ΕΚΤ του τραπεζικού της συστήματος εάν αυτή η συνολική αξιολόγηση, η σφαιρική αξιολόγηση εντοπίσει κάποιες αδυναμίες, κάποια σημεία ευάλωτα, θα πρέπει η χώρα αυτή να φέρει πέρα σε κάποιες δράσεις, μεταξύ των οποίων μάλλον πάνω στις από τις οποίες θα κρυθεί, από την υλοποίησή τους θα κρυθεί η συμφωνία στενή συνεργασία. Από την άλλη, το να μπει κανεί σε μια νομισματική ένωση με τραπεζικές αδυναμίες και έφτραστα σημεία, σίγουρα δεν είναι κάτι το λογικό. Ευχαριστούμε Πέντρο Σίλβα Περέιρα από τους Σοσιαλιστές και δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, όπως και άλλοι και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε βεβαίως ε, συμβατά με την εντολή που είχατε να σώσετε τον ευρώ, το ευρώ και αυτά τα είναι πολύ σημαντικά και όχι, όχι μόνο σας συγχαίρω γιατί ήσασταν ε, ε, σοφός αλλά και γιατί είχατε την αποφασιστικότητα να αντιδράσετε σε διαφωνίες μέσα στο Συμβούλιο και εκτός Συμβουλίου. Για άλλη μια φορά χαιρετίζω τα νέα επεκτατικά μέτρα που ανακοινώσατε, αλλά βλέπουμε και πάλι αντίσταση να υπάρχει. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι κάποια μέλη ε, του ε, Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ήδη ε, κάνει δηλώσεις κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν και συμφωνείτε ότι θα ήταν ίσως καλύτερα να υπάρχει περισσότερη αλληλεγγύη μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, ε, το μήνυμά σας υπέρ μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικό. Ε, ζητάτε να υπάρχει επεκτατική πολιτική από τις χώρες που έχουν τέτοιο δημοσιονομικό χώρο, αλλά φαίνεται ότι το μήνυμα δεν είναι πια ένα μήνυμα που εκπέμπεται προς την Γερμανία ή την Ολλανδία. Συμφωνείτε λοιπόν ότι οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για επεκτατική πολιτική ότι είναι περισσότερες πια αυτές οι χώρες και τώρα έχουμε πλέον τις ε, προϋποθέσεις ε, για ε, πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στις χώρες της Ευρωζώνης. Λοιπόν, να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, οι διαφωνίες στην πολιτική είναι συνηθισμένες. Αν δείτε την τελευταία απόφαση που λήφθη από το Ομοσπονδική Τράπεζα των ΗΠΑ, ελήφθη με διαφωνούσα μειονότητα. Ακόμα και αυτοί που διαφώνησαν, διαφώνησαν ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικές φορές ήθιστε ορισμένες από αυτές τις διαφωνίες να δημοσιοποιούνται. Ε, μην ξεχνάτε ότι εγώ στους, ε, στα έξι μου χρόνια ε, το έζησα αυτό όταν ήμουν ε, κεντρικός τραπεζής στην Ιταλία και ο κύριος Τρισέ και αυτό στη Γαλλία το έζησε και αυτός. Εγώ δεν θυμάμαι ε, ποτέ να είπα κάτι για τη νομισματική πολιτική που να ήταν αντίθετο σε αυτά που αποφάσισε η ΕΚΤ. Μπας περιπτώσει, ε, η μορφή με την οποία δημοσιοποιείται η διαφωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική κυρίως ε, όταν έχουμε μία ένωση νομισματική που εφαρμόζεται από πολλέ χώρε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει σύνεση έτσι ώστε να μην υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των αποφάσεών μας. Αυτό το σχόλιο έχω μόνο να κάνω. Για τη δεύτερη ερώτησή σα για τη δημοσιονομική πολιτική, εναπόκειται στην Επιτροπή και στους κανόνες ε, το κατά πόσον ε, θα αναθεωρηθεί η δημοσιονομική πολιτική ε, στο μέλλον. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω, να ονοματίσω χώρες που έχουν δημοσιονομικό χώρο. Η εξέταση γίνεται με βάση τους υπάρχοντες κανόνες και με βάση το πώς ερμηνεύει κανείς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχουμε χώρες με υψηλά χρέη που θα πρέπει να είναι συνετές και άλλες ε, που έχουν δημοσιονομικό χώρο θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικές. Αλλά σας είπα, όλα αυτά ενδεχομένως θα αναθεωρηθούν και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι κανόνες θα αναπροσδιοριστούν, θα είναι αποτελεσματικοί και λογικοί. Ευχαριστώ. Τσικλίνιας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έρχομαι από τη Λιθουανία, μια μικρή χώρα που προσπάθησε και αυτή να αντιμετωπίσει την κρίση όταν μας ε, χτύπησε βαριά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα επαγγελματικά σας και πολύ επαγγελματικά σχόλια βασικά που μας κάνετε εδώ. Θέλω να, να σχολιάσω Αυτά που είπε ο Κλώδιο Μπάριο και αν Μπασάνλη όσον αφορά τις ε, τραπεζικές συνονίες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τις απόψεις σας. Λένε ότι το ωφέλη και το κόστος, ο συνδυασμός αυτός επιδεινώνεται. Και τι μπορεί να κάνει νομισματική πολιτική γι' αυτό. Και το δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι τα μέτρα, τα μη συμβατικά μέτρα, είναι έκτακτα για να αντιμετωπιστούν πολύ ιδιαίτερε συνθήκες. Τώρα εσείς αναφερθήκατε στις παρενέργειες. Αρνητικές συνέπειες τέτοιων μέτρων που ε, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν αποταμιεύουν ε, το ίδιο πρόθυμα. Αναφερθήκατε επίσης στις δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας. Αλλά εδώ μπαίνουμε αν θέλετε, στη δημοσιονομική πτυχή, δηλαδή την πολιτική. Δεν είναι και αυτό μια παρενέργεια. Έπειτα η έξοδος από τα μη συμβατικά μέτρα είναι κάτι εφικτό. Τώρα εσείς που θα αποχωρήσετε δεν είναι πολύ επικίνδυνη η ισορροπία αυτή των αρνητικών ε, επιτοκίων με τις προσδοκίες που δημιουργούνται από πλευρά των επιχειρήσεων ε, και του κοινού γενικότερα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει απόδειξη ότι αυξάνονται οι αποταμιεύσεις με αρνητικά επιτόκια. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει καμιά απόδειξη ότι οι τράπεζες μειώνουν τον δανεισμό ως συνέπεια αρνητικών επιτοκίων στις, ε, στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεως, καταθέσεις δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και το αντίστροφο. Το δεύτερο είναι πότε θα βγούμε από αυτά τα μέτρα. Ε, θα βγούμε όταν η οικονομία βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε μία έξοδος να μην δημιουργήσει συστολή στην ίδια την οικονομία. Και αν πάμε πίσω ε, τέλη 2017 αρχές 2018 υπήρξε μια αύξηση κάτι το οποίο έδειχνε ότι προχωράμε προς μια τέτοια έξοδο από αυτήν την ιδιαίτερα διευκολυντική οικονομική ε, πολιτική, νομισματική πολιτική. Οπότε αυτό είναι το κλειδί. Να είμαστε σε θέση να πάρουμε κάποια μέτρα κανονικοποίησης, χωρίς όμως να δυσκολεύουμε τις οικονομικές συνθήκες, γιατί συνοδεύονται από βελτίωση της οικονομίας. Θα θυμόσαστε τι είπα στη Σύντρα τον Ιούνιο του 2017, που ήταν ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Όπως είπα και στην αρχή, βλέπουμε μια προοπτική σταδημιακά επιδίνωσης και με διακοπές, αλλά και πάλι έρχομαι στην δημοσιονομική πολιτική. Αν παρέμβει η δημοσιονομική πολιτική και βοηθήσει, τότε σίγουρα η νομισματική πολιτική θα έχει πιο ελαφρύ ρόλο. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα θα συνεχίσει να λειτουργεί η νομισματική πολιτική και θα παρακολουθεί τις παρενέργειες αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Μπέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου ξεπέρασαν λίγο το χρόνο του. Ελπίζω ότι θα μεταχειριστείτε με την ίδια επίκαια. Εδώ κρατάω μια φράουλα. Και σύμφωνα με το ζωγράφο Ερώνυμο Μπός, είναι ε, σύμβολο της επίγειας απόλαυσης και ειδονής η φράουλα. Κάποιοι το λένε αυτό για την ποσοτική χαλάρωση επίσης. Και τώρα θα συνεχίσω στα γερμανικά. Χαίρετε, Πρόεδρε. Γεια σας. Το 2011, μάλλον από το 2011, τυπώσατε περισσότερα χρήματα και παραβιάσατε περισσότερους κανόνες από οποιονδήποτε, οποτεδήποτε στην ιστορία. Και ακόμα και η κυρία Λαγκάρτ το ομολόγησε αυτό όταν ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Παρόλα αυτά, από το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανεπτύχθη με τον ίδιο ρυθμό όπως ο υπόλοιπο κόσμος, ε, εξαιρουμένης βέβαια της Ιαπωνίας και η Ευρωζώνη ακόμα λιγότερο από τις υπόλοιπε ζώνες. Η δική σας ε, η νομισματική πολιτική είναι μια πολιτική αποτυχίας ε, για πάρα πολλά κράτη. Αυτό είναι προγραμματισμένο και ίσως να μην μπορούμε να το φανταστούμε στην απόλυτη έκτασή του. Στην συνέντευξη που δώσατε είπατε ότι τα αίτια όλων αυτών είναι η παγκόσμια οικονομία, η εμπορική πόλεμη και το Brexit. Επειδή όμως όλα αυτά μάλλον δεν βοηθούν, για το λόγο αυτό χορηγήσατε στο ευρώ διπλάσια δόση φαρμάκου, παρότι γνωρίζουμε ότι η ποσοτική χαλάρωση το μόνο που θα επιτύχει είναι να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους ε, φτωχούς φτωχότερους. Ο συμπατριώτης σας, ο κύριος Μακιαβέλη είπε ότι η επιτυχία μας και η αποτυχία μας κατά το ίμιση οφείλονται στην μοίρα μας. Το υπόλοιπο ίμιση αφορά την θεά της τύχης, τη φορτούνα. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, μήπως ε, δεν κάνετε τη ζωή πολύ εύκολη με το να αποδίδετε στη φορτούνα, τη θεά της τύχης, όλη αυτή την υποτυχία και την εξατλίωση. Γιατί σε τελική ανάλυση η παγκόσμια οικονομία αφορά όλους όλους τους πολίτες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. No, no, we are not blaming fortune. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τη θεά τύχη. Μην ανησυχείτε. Αλλά να πω αρχικώς ότι η κυρία Λαγκάρντ δεν είπε ότι οι δράσεις της νομισματικής πολιτικής ήταν παραβίαση της συνθήκης τα συμβατικά και ασυμβατικά μέτρα που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλα έγιναν στα πλαίσια της επιδίωξης σταθεροποίησης των τιμών στόχο που προβλέπεται από το καταστατικό τη. Όπω είπα επανειλημμένω σήμερα, κάποιε φορέ χρειάστηκαν αντισυμβατικά ε, πολιτικά μέτρα για να έχουμε περαιτέρω ε, αντιμετώπιση των ε, κινδύνων και των πιέσεων. Και φτάσαμε στα όρια των δυνατοτήτων μας. Κάποιες φορές είχαμε τα ομόλογα σε ευθεροχές αγορές ως μέτρο και αυτό εξυπηρέτησε, όπως φάνηκε πριν από λίγα λεπτά, αυτό εξυπηρέτησε στο να φτάσουμε το στόχο της σύγκλησης ή τις, τους στόχους για τον πληθωρισμό τους, μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον. Τα εργαλεία αυτά σεβάστηκαν τα όρια και τα σύνορα της εντολής μας. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δύο αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, για τις απευθείας ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και μετά για τον δημόσιο τομέα και τις σχετικές αγορές. Το ίδιο το δικαστήριο επανεπιβεβαίωσε την αναλογικότητα των μέτρων αυτών. Δηλαδή, τα μέτρα αυτά ήταν ακριβώς τα μέτρα που χρειάζονταν υπό τις δεδομένες συνθήκες και σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους της νομισματικής πολιτικής. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ΕΚΤ χρησιμοποίησε τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να πετύχει τους νόμιμους και θεμητούς στόχους στο βαθμό που ήταν αναλογικός ως προς τις ανάγκες διόρθωσης των ελλείψεων στην πολιτική του πληθωρισμού και την ικανοποίηση των αναγκών της σταθεροποίησης των τιμών. Ταυτόχρονα με τις αγορές των κρατικών ομολόγων βάσει του σχετικού προγράμματος, και αυτά ήταν συμβατά με την απαγόρευση της ε, μακροοικονομικής χρηματοδότησης, όπως ορίζει το άρθρο 1 στο εδάφιο 2 υπό εδάφιο 3 της συνθήκης. Νομίζω απήντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γιούτσικα, για την Γιούτσικα από τους εταιρετικούς και μεταρρυθμιστές. Μάλλον εγώ είμαι. Με συγχωρείτε για την κακή προφορά. Και εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον της ζωής σας κύριε Ντράγκη. Δύο ερωτήσεις για τον ισολογισμό της ΕΚΤ. Έχει διπλασιαστεί σε δύο χρόνια περίπου 40% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3 δις ευρώ. Βλέπετε κανένα κίνδυνο σε αυτή την τεράστια διόγκωση Και η δεύτερη ερώτηση. Γιατί η ΕΚΤ δεν έδωσε στο ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες όπως ζητήθηκε για να μπορέσουμε να δούμε την εποπτεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών εμένα μου φαίνεται ότι αυτό κάπως έπληξε την αξιοπιστία της ΕΚΤ. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση συμφωνώ, δεδομένου του όγκου των επιπέδων που έχει φτάσει ο ισολογισμός, παρακολουθούμε όλους τους ενδεχόμενους παρελκόμενους κινδύνους. Τι μπορεί να προκαλέσουν οι αλλαγές στα επιτόκια, ας πούμε, στον ισολογισμό της ΕΚΤ. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους στην αγορά, ο ισολογισμός της ΕΚΤ δεν είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς των επικοινωνιών απευθείας, διότι αξιολογείται με βάση το επίπεδο απόσβεσης και αποπληρωμής του, του χρέους και όχι με βάση όρους της αγοράς. Έχουμε πολλά όπλα κατά των συστημικών κινδύνων, κατά των εμπορικών κινδύνων. Μια σειρά από διατάξεις και περιπτώσεις που δεν τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή, είναι πολύ άριθμες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον κίνδυνο από τις πιστώσεις. Α, τον κίνδυνο από τις αγορές. Να προσθέσω ότι όταν πηγαίνουμε στα παράγωγα, στις εγγυήσει, που είναι επίσης ένα μέρος της δουλειάς της ε, ΕΚΤ, υπάρχουν κριτήρια ρεσιμότητας. Παρόλο που οι κανόνες για τις εγγυήσει άλλαξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα κριτήρια ρεσιμότητας είναι ακόμα πολύ υψηλό επίπεδο και έγιναν και κουρέματα, όπως ξέρετε, για τον ίδιο σκοπό. Γι' αυτό έχουμε και μια υπηρεσία παρακολούθησης του κινδύνου και μάλιστα πολύ καλά επανδρομένη και επιγυναικωμένη στην ΕΚ. Αλλά για το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σίγουρα έχει φωτιστεί πολύ σωστά η σχέση μεταξύ ΕΚΤ στην νομισματική της λειτουργία και της ΕΚΤ ως ε, παράγοντα αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως το βασικό σημείο τώρα, το βασικό σημείο νομίζω το έχει απαντήσει κιόλα η διάσταση της νομισματικής ένωσης. Αλλά αλλά πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών βάσει της απόφασης του δικαστηρίου, παρόλο που έχει καλυφθεί αυτό από το μνημόνιο συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εύα Μαϊντό, ΕΛΚ. Πρόεδρε, χαίρομαι που είσαστε μαζί μας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τους συναδέρφους και να πω και εγώ ότι η ΕΚΤ είναι ισχυρότερη, βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση. Πάντως εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προλαμβάνει τις κρίσεις πολύ περισσότερο από ότι να τις διαχειρίζεται. Και νομίζω ότι κάποιες από τις τελευταίες πολιτικές που υλοποίησατε ακριβώς αυτό προσπαθούν να κάνουν. Τώρα το θέμα των επιτοκίων η πολιτική σας απέναντι στα επιτόκια έχει φτάσει στα ωριά της, πιστεύω. Και με αναρωτιέται ο κόσμος κατά πόσο τελικά μπορεί η έκτη με τα μέτρα αυτά να επηρεάσει σημαντικά τον, ε, τα επιτόκια. Θα έλεγα λοιπόν, να τώρα βρισκόσαστε στο τέλος αυτής της επιτυχούς εντολής σας. Τι άλλες εξουσίες πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει έκτη για να μπορέσει να διασφαλίσει ακόμα καλύτερα ε, το ευρώ και να εγγυθεί τη σταθερότητα τιμών ή τι εξουσίες θα θέλετε να είχε η ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας. Τώρα δεν άκουσα τους συναδέρφους να ρωτάνε για το Brexit. Ε, πλησιάζουμε από ό,τι φαίνεται και ε, σίγουρα η νομοθεσία ε, για την ε, Τραπεζική Ένωση και τα λοιπά θα μπορούσε να εφαρμόζεται στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα υπάρξουν ίσως διαφορές στην, στο προληπτικό σκέλος, στο εποπτικό σκέλος. Αν τελικά μέσα σε επόμενες εβδομάδες υλοποιηθεί το Brexit, ποια είναι η γνώση σας. και ό,τι σκέψεις έχετε για την περίοδο μετά, κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ε, δημοσιονομική πολιτική, τι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα καλύτερα οι κυβερνήσεις. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε για το Brexit, δεν κατάλαβα, και την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συγγνώμη. Είναι προετοιμασμένη η ΕΚΤ για την περίπτωση να μην υπάρξει συμφωνία για τον Brexit. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Απάντηση. Ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ μαζί σας για αυτά που είπατε όσον αφορά τη φύση των πρόσφατων μέτρων μας. Εμείς αντιδρούμε ε, σε μια καθοδική πορεία προπτικής. Δεν αντιδρούμε δηλαδή σε κάτι το οποίο έχει ήδη λάβει χώρα, αλλά στην προπτική του να λάβει χώρα. Και η κατάσταση είναι σχετικά καλή και αυτό μας δίνει εμπιστοσύνη ότι τελικά αν δράσουμε τώρα θα υπάρξει σύγκληση του πληθωρισμού προς το στόχο. Τώρα με ρωτάτε τι άλλες εξουσίες θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα αν δείτε τώρα τις εξουσίες μας, είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν οι περισσότερες ε, κεντρικές ε, τράπεζες σε εξίσου μεγάλες δικαιοδοσίες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η ΕΚΤ την εργαλειοθήκη της. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ε, στις δυσκολίες, πάντα βέβαια σύμφωνα με την εντολή της και το στόχο που είναι η σταθερότητα τιμών. Τώρα, κατά πόσο οι πολιτικέ μα είναι αποτελεσματικές ή όχι, εμείς πιστεύουμε και το είπα πριν από λίγο, ότι συσσωρευτικά η απάντησή μας οδήγησε σε ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως κατά πόσο είναι αποτελεσματικές ή όχι είναι ένα ανοιχτό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε όλες τις κεντρικέ τράπεζε του κόσμου. Τώρα είμαστε σε ένα κόσμο μεγάλης ρευστότητας παντού, λίγο πολύ εξίσου επεκτατικές νομισματικές πολιτικές ακολουθούνται από όλες τις κεντρικές τράπεζες, αν δείτε τα επιχειρήματα και την πολεμική που ακούγεται για διάφορες αποφάσεις μας, θα πείτε ότι είναι έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στην Ευρώπη μόνο. Όμως δεν ισχύει αυτό. Λίγο πολύ το ίδιο γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς, το ερώτημα το κατά πόσο αυτή η νομισματική πολιτική έχει φτάσει στα όρια της ή όχι είναι ένα γενικό ερώτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ακόμα αποτελεσματική. Ε, βέβαια, οι δευτερεύουσες συνέπειες και λοιπά είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Εξού και η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να συμπληρώνει την νομισματική πολιτική. Είναι κάτι το οποίο ισχύει όμως και σε άλλες δικαιοδοσίες. Και βλέπετε τις διαφορές όσον αφορά και τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Και οι συνολικοί παράγοντες οι οποίοι ε, περιορίζουν τις ε, προοπτικές, τις πληθωριστικές κτλ. ισχύουν και αλλού. Και δεν ισχύουν μόνο στην Ευρωζώνη. Τώρα για το Brexit. Η ΕΚΤ με την Τράπεζα της Αγγλίας τρία χρόνια τώρα συνεργάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα πρόπτα και φυσικά ένα Brexit χωρίς συμφωνία είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι πολύ βασικό αυτό που έχουμε πει για τις προσωρινές ισοτιμίες και έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται και ιδιωτικό τομέας προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να παρακολουθούμε τις δικές τους δράσεις. Τώρα, κατά πόσο ο ιδιωτικό τομέας θα αναλάβει όλο τον κίνδυνο ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Ε, συχνά ο κόσμος λέει όχι, ότι δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος. Έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον, ώστε να εκφραστεί ποσοτικά δηλαδή. Μπίλι Κέλεχερ από το Renew Europe. ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω, κύριε Ντράγκη. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω ότι εσείς ε, το όνομά σας έχει αφήσει ιστορία στη χώρα μας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά ε, το σύμφωνο σταθερότητας, ε, μιλάμε για την ανάπτυξη και για τα ελλείμματα. Πώς ακριβώς μπορείτε να δώσετε κίνητρα στις ε, κυβερνήσεις έτσι ώστε να κινούνται αντικυκλικά. Με άλλα λόγια, οι χώρες μπορούν να δαπανίσουν μόνο όταν έχουν χρήματα και όταν χρειάζονται να δαπανίσουν δεν έχουν χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορείτε να δώσετε κίνητρα στις οικονομίες και αναφέρομαι κυρίως στην Γερμανία. Γιατί η Γερμανία ε, δεν αρχίζει να δαπανά και οι ε, εξαγωγές της να είναι πιο προστές ε, για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, Τραπεζικής Ένωσης ε, και του νέου εποπτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο καιρό αναφέρθηκε ότι ίσως περιοριστούν ε, οι πρακτικές δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόσφατα μιλήσατε στην Ιρλανδία σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου είπατε ότι οι Ιρλανδικές τράπεζες λειτουργούν σχεδόν μονοπωλιακά, ιονή μονοπωλιακά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δάνεια που να χορηγούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς λόγω των περισμών που υπάρχουν. Και ε, κατά τα άλλα, μήπως έχουμε μια κατάσταση όπου στην Ιρλανδία, όπου προσπαθούν ε, να ανακτήσουν τα κέρδη τους ε, περισσότερο με υπερβολικά επιτόκια και όχι δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λοιπόν, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, όπως είπα και προηγουμένως, η εμπειρία που έχουμε κάνει είναι ότι οι κανόνες είναι αποτελεσματικοί ε, στο να περιορίσουν το χρέος. Ε, ως εκ τούτου οι κανόνες είναι λογικοί, αλλά πια ε, πλέον δεν είναι αποτελεσματικοί. Και έτσι πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση που κάνατε. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αισιόδοξο ότι η Κομισιόν και η ΕΚΤ θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Όταν λοιπόν μιλάμε για δαπάνες, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι ακριβώς δαπάνες έχουμε κατά νου. Και είναι απόλυτα σαφές ότι ακόμα και σε χώρες που έχουν δημοσιονομικό χώρο, οι δαπάνες που γίνονται θα πρέπει να είναι οι δαπάνες που ενισχύουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης, δηλαδή παραγωγικότητα, άρα δηλαδή δαπάνες να γίνονται στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στην πληροφορική, στην παιδεία. Αυτά ενισχύουν ε, μακροπρόθεσμα τις δυνατότητες μιας χώρας και Νομίζω έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι δικές σας επιφυλάξεις του να γίνονται οι εξαγωγές πιο αποτελεσματικές. Θα γίνουν πιο αποτελεσματικές, είναι τεχνολογικά πιο προχωρημένες και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Το να αναθεωρούν τον προπολογισμό τους ε, με έναν τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη, αυτό είναι το κλειδί της όλης ιστορίας. Το δεύτερο που άκουσα να εκφράζεται πολλές φορές είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγεί σε μείωση του δανεισμού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε τέτοιου είδους ενδείξεις. Έχουμε να το πω Έχουμε ενδείξεις ε, ότι αυξάνεται ο δανεισμός, και προς τα νοικοκυριά και προς τις επιχειρήσεις. Βέβαια εξαρτάται ε, σε μεγάλο βαθμό από ποιες επιχειρήσεις και σε ποιες χώρες. Και σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι δεν υπάρχει περιορισμός του δανεισμού προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν θυμάμαι καλά, ε, τα spread δανεισμού ανάμεσα σε ε, μάλλον η διαφορά, το, η απόσταση δανεισμού ανάμεσα μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις έχει περιοριστεί, το χάσμα του δανεισμού. Όμως, αν τελικά η Τραπεζική Ένωση σημαίνει μεγαλύτερα ποσά, ε, διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί έχουμε οικονομίες κλίμακας και πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Αυτά συνεπάγονται και αρνητικά όπως είναι ότι θα γνούνται λιγάκι οι μικροί πελάτες. Και υπάρχει ένας άλλος τομέας ε, που είναι διαφορετικός. Εκεί πρόκειται για τις ε, απαιτήσεις της Συμφωνίας Βασιλεία 3 που ζητάνε κεφαλαϊκή εξασφάλιση έναντι επιχειρήσεων που έχουν ιστορικό υψηλού κινδύνου. Ε, και αν μπορεί να υπάρξει κάποιος περισμός δανεισμού είναι από αυτό, από τη Βασιλεία 3 και όχι τόσο από τις ίδιες τις τράπεζες. Ο κύριο Πεντιτσίνη, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσά Πρόεδρε Ντράγκη που είστε εδώ για να απαντήσετε στι ερωτήσει μα. Πρώτα απ' όλα, μιλήσατε επανειλημμένω για διαφορετικέ μεταρρυθμίσει διαφορετικών χωρών. Όμω δεν μιλήσατε για διευθυντικέ μεταρρυθμίσει τη Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι αυτό είναι θέμα απόφαση των πολιτικών. Συμφωνώ. Όμω, εμεί οι πολιτικοί, εμεί που είμαστε πολιτικοί ηθήνοντε, χρειαζόμαστε και μια τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και το κύρο το δικό σα για να μπορούμε να χαράξουμε καλύτερα τι πολιτικέ μα αποφάσει. Επανειλημμένω γίνεται λόγο για τι χώρε που δεν είναι καλοί μαθητέ, που δεν κάναν τα μαθήματά του. Όμω, τι υπονοείται με αυτό. Μιλάτε για τις χώρες με ψηλό χρέος όπως η Ιταλία, διότι ο συνάδελφος ε, Γκερτάνο το σχολίασε προηγουμένως. Ίσως να μην γνωρίζουν όλοι ότι η Ιταλία από το 1992 καταγράφει πρωτογενή ανάπτυξη. Και αυτό σημαίνει ότι οι φόροι που πληρώνει η Ιταλία είναι πολύ υψηλότερη από το δημόσιο χρέο. Η διαφορά είναι ότι περίπου 30 δις το χρόνο. Εμεί κάνουμε λοιπόν τα μαθήματά μα σωστά, είμαστε καλοί μαθητέ. Όμω, προκύπτει να είναι αρνητικό το ΕΠ, διότι α, αυτά που πληρώνουμε ω το δημόσιο χρέο είναι διπλάσιο από το πρωτογενές κέρδο. Ω τώρα έχουμε πληρώσει επιτόκια για το δημόσιο χρέο, διπλάσια από το ίδιο το χρέο. Ποιο από εσά θα συνέκρινε ένα αμάξι των 10.000 ευρώ και θα πλήρωνε γι' αυτό τόκους 30.000 ευρώ. Είναι τεράστια ειδικία. Και πρέπει να κάνουμε σωστά για τους λογαριασμούς. Πρέπει να κάνουμε εδώ μια διάκριση. Πού είναι το πραγματικό συμφέρον και πού η κερδοσκοπία. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στις χρηματαγορές που πραγματικά παίρνουν τόκους τοκογλυφικούς από κάποια κράτη όταν αγοράζουν χρέος εδώ λοιπόν, ποια είναι η δική σα άποψη για το γεγονό ότι η ΕΚΤ πρέπει εδώ να έχει και ένα ρόλο. Ένα ρόλο που να τη επιτρέπει να παρέμβει στην πρωτογενή αγορά και να ορίσει ένα τόκο για τα κρατικά ομόλογα κατώτερο ή τα κρατικά αξιόγραφα κατώτερο από το επίπεδο του πληθωρισμού ή να είναι, μάλλον αν ήταν υψηλότερο το επίπεδο του πληθωρισμού από τα κρατικά ομόλογα, θα, θα μπορούσαν να κερδίσουν τα κράτη από την πώληση ομολόγων χωρί να καταστραφούν με πολιτικέ λιτότητε οι χώρε μα όπω ε, η Ιταλική αγορά, α πούμε. Θα πω Πρώτα απ' όλα κάτι στα Ιταλικά. Δεν προβλέπεται από τη συνθήκη ή από το καταστατικό τη ΕΚΤ ούτε από τι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Η ΕΚΤ έχει ω στόχο την σταθεροποίηση των τιμών και όχι τη χρηματοδότηση των ε, χρεών των επιμέρου χωρών. Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορούμε εμεί να παρέμβουμε στους τόκου και στα επιτόκια των επιμέρου χωρών. Δεν το επιτρέπουν οι συνθήκε ή το καταστατικό της ΕΚΤ ε, ή οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Ο στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθεροποίηση των τιμών και όχι η χρηματοδότηση χρεών και δημοσιονομικών ελλημάτων χωρών. Αν αλλάξετε τη συνθήκη, θα το κάνουμε αυτό που μας ζητάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λούωμα, σοσιαλιστές και δημοκράτες. δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου, όπως και άλλοι που σέβονται το έργο σας κύριε Ντράγκη, να σας ευχαριστήσω. Εγώ έρχομαι από μια πολύ βόρεια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όνομά σας πάντα συνδέεται με μια επιτυχή νομισματική πολιτική και με τη διάσωση του ευρώ και της ευρωζώνης. Έχω δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την εντολή σας και τη θητεία σα. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τον πληθωρισμό και η δεύτερη έχει να κάνει με τους κανόνες τη οικονομική και Νομισματικής Ένωση. Για τον πληθωρισμό πρώτα απ' όλα. Περιμένουμε ακόμα, όπως και παλιά, όταν ο πληθωρισμός ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα ή μήπω στην εποχή της παγκοσμιοποίηση, ο κίνδυνος υψηλού πληθωρισμού είναι χαμηλότερος από ό,τι κατά το παρελθόν και ο κίνδυνο για την απασχόληση είναι μεγαλύτερος από ό,τι κατά το παρελθόν. Και χαίρομαι που όταν μιλήσατε για τους κανόνες της ΙΟΝΕ είπατε ότι χρειάζονται αλλαγές ότι δεν κάνουμε πλέον προκυκλικές πολιτικές. Οι κανόνες όμως που έχουμε λένε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε χρέος. Όταν όμως υπάρχει υπερβολική ρευστότητα, δεν έχουμε κανόνες για το τι να κάνουμε, ούτε έχουμε κανόνες για τις χώρες εκείνες που τα πηγαίνουν καλά. Πώς θα μπορούσαν εκείνες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο προς όφελος ολόκληρης της Ευρωζώνης. Απάντηση. Πιστεύω ότι η απάντηση στην ερώτησή σας έχει να κάνει με μια κεντρική ε, δημοσιονομική ικανότητα. Ένα δηλαδή δημοσιονομικό μέσο το οποίο να βοηθάει στην σταθεροποίηση του οικονομικού κύκλου παντού στην Ευρωζώνη για διάφορες χώρες μέλη. Τώρα, είπα και πριν ότι για να είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο δημοσιονομικό εργαλείο πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος και πρέπει να λειτουργεί αυτόματα και έγκαιρα. Αλλά για να έχουμε αυτήν τη δημοσιονομική ικανότητα πρέπει να στηριχτούμε από όλες τις χώρες μέλη. Και νομίζω αυτό ακριβώς ρωτάτε. Με ποιο τρόπο δηλαδή η αλληλεγγύη παρεμβαίνει από όλες τις χώρες. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από ε, υπευθυνότητα, από την ευθύνη που αναλαμβάνουν ε, κάποιες χώρες. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συμφωνήσουμε για αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα. Άπαξ και το έχουμε, εντάξει, είναι πολύ λογικό, έχει νόημα, αλλά συγχρόνως πρέπει να ξεπεράσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης που ίσως υπάρχει σε διάφορες χώρες για την υπευθυνότητα με την οποία ε, ασκούν την ε, δημοσιονομική τους πολιτική. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρόεδρος. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι σήμερα. Ε, συγγνώμη, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Πρέπει να περάσουμε ευθύ αμέσω στο επόμενο θέμα. Οπότε, κύριε Ντράγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον νομισματικό διάλογο. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 4, που είναι η ακρόαση Και καλωσορίζω εδώ και πάλι τον κύριο Ντράγκη υπό την ιδιότητά του του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική πολιτική. Έχουμε τους ίδιους κανόνες που είχαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Τέσσερα λεπτά αναερώτηση γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Οπότε παρακαλώ κύριε Ντράγκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου να απευθύνομαι στην Επιτροπή σα για δεύτερη φορά φέτο. Είναι η τελευταία μου προσέλευση στο Ευρωκοινοβούλιο από την ιδιότητά μου ω Προέδρου του ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, αλλά είναι η πρώτη στην ένατη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου. Την τελευταία φορά που μίλησα στην Επιτροπή σα ω πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, συζήτησα τα όσα είχαμε πετύχει στα επίπεδα τη μακροπροληπτική πολιτική για τι βασικέ προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Σήμερα θα ήθελα να θίξω το θέμα τη αγορά ακινήτων, ε, πράγμα που το Συμβούλιο μα έχει μελετήσει ω μέρο τη τακτική διαδικασία παρακολούθηση του τι συμβαίνει στι χώρε μέλη. Όπω έχουμε συζητήσει επανειλημμένω προ το παρελθόν με την Επιτροπή σας, σα, οι εξελίξει στην αγορά των ακινήτων μπορεί να έχουν σοβαρότατε επιπτώσει για την ε, οικονομική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία το να βεβαιωθούμε ότι η Επιτροπή σας γνωρίζει πλήρως τις απόψεις σχετικά του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είναι σημαντικό ε, τμήμα της υποχρέωσης λογοδοσίας που έχουμε προς το Ευρωκοινοβούλιο. Το Συμβούλιο μας ιδρύθηκε για να παρακολουθεί τους κινδύνους προς την ε, οικονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβλέπει κατάλληλες πολιτικές αντιδράσεις. Έπρεπε να ασκείται πίεση από μοτίμους και να αντιμετωπίσουμε και την ε, διάθεση για αδράνεια, την ε, ροπή προ την αδράνεια που υπήρχε. Γι' αυτό υπάρχουν προειδοποιήσει και εντοπίζουμε ευάλωτα σημεία και τάσει που μπορεί να πλήξουν την οικονομική σταθερότητα. Πρέπει όμω να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και πολλέ φορέ να εκδώσουμε συστάσει που όχι μόνο εντοπίζουν κινδύνου, αλλά στοχεύουν και την ανάλογη δράση προ αποκατάσταση. Με βάση λοιπόν τη μακροπρόθεσμη ανάλυση του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στον, ε, στην αγορά κινήτων, το Συμβούλιο μα αυτή τη στιγμή εξέδωσε πέντε σημεία προειδοποίηση και έξι συστάσει σε σχέση με μακροπρόθεσμα σημεία ευπάθεια στον τομέα αυτό. Η μεθοδολογία και η ανάλυση που υπόκεινται ε, και στηρίζουν τις αποφάσεις μας τεκμηριώνονται από τρεις ε, εκθέσεις. Οι προειδοποιήσει και οι συστάσεις ε, αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά και έχουν να κάνουν και με τα εργαλεία που διατίθενται στι επιμέρου χώρε, την εφαρμογή του και διάφορο, του διάφορου συσχετισμού μεταξύ των ευάλωτων σημείων, των σημείων ευπάθεια. Τα σημεία αυτά επάθεια μπορεί να έχουν να κάνουν με το χρέο των οικοκυριών, την ε, ε, αύξηση των δανείων τους, ε, τις προδιαγραφές για το δανεισμό ή τις αλλαγές στις τιμές στην αγορά κινήτων. Τα εργαλεία μακροληπτικής ε, πρόληψης μπορεί να αντιμετωπιστούν εφόσον χρησιμοποιούν τα νομικά εργαλεία που διαθέτουμε. Η τις αλλαγες στις τιμες στην αγορα κινητων τα εργαλεια μακρολεπτικης προληψης μπορει να αντιμετωπιστουν εφοσον χρησιμοποιουν τα νομικα εργαλεια που διαθετουμε η αναλυση μας δείχνει ότι σε κάποιες χώρες οι αρχές δεν έχουν αρκετά εργαλεία που να βασίζονται στην ε, πλευρά του δανειστή ενώ κάποιες άλλες χώρες μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν άλλα περισσότερα εργαλεία που διατίθεται. Πρέπει να σημειώσω ότι ε, από την τελευταία φορά που ήρθα εδώ έχουμε εκδώσει την ετήσια έκθεσή μας που περιγράφει την ανάλυση κινδύνου και τις συνεισφορές μας για το πλαίσιο μακροπολιτικής ε, πολιτικής από την 1η Απριλίου 2018 στην 31η Μαρτίου 2019. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η δουλειά μα στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου σε επίπεδο τεχνοκρατικό θα συζητηθεί σύντομα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε τρει μέρε θα ανταλλάξουμε απόψει για τη μακροπροληπτική χρήση των ε, περιθωρίων και των ε, κουρεμάτων, μέρο τη στρατηγική μα για να έχουμε μια καλύτερη εργαλειοθήκη μακροπολιτική ε, πολιτική. Επίση, θα δούμε πώ θα έχουμε ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτών από τι χώρε υποδοχή και χώρε προέλευση και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία των επιμέρου χρηματοποιητών θα συνεχίσουμε να αναλύουμε και τις επιπτώσεις των κυβερνοκινδύνων για την οικονομική σταθερότητα και γενικότερα θα συνεχίσουμε να μελετούμε πώ μπορούμε να αλλάξουμε την διάρθρωση του χρηματοοικονομικού μα συστήματο, τον ρόλο που μπορεί να παίζουν τα τεστ για κόπωση ή ελέγχου των πιέσεων και του τι περαιτέρω έχουμε αποκομίσει ε, ως προς τη μακροπολιτική πολιτική. Η τέταρτη ετήσια διασκεψή μας ξεκινά την Πέμπτη και προσκαλώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής σας να πάρουν μέρος στην διάσκεψη αυτή στη Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank you. Uh, now we have Georgios. Uh, Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κίτσος τώρα από το Ε, πρόεδρε Ντράγκη, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συμβολή σας στην ενίσχυση του ευρώ και την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και φυσικά για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, θέλω να σας θέσω ερωτήματα για το ελληνικό συστημικό ρίσκο στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Πρώτον, είμαστε πλέον σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ακόμη και για χώρες με υπερβολικό χρέος όπως η Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τις παραδοχές για υψηλά επιτόκια στις μελέτες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και να κάνουμε υπολογισμούς με χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλότερο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να μειώσουμε τα μελλοντικά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή όχι. Δεύτερον, θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών γιατί είναι σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρωζώνη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο φιλική για την οικονομία. Πώς εκτιμάτε ότι εξελίσσεται η κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τρίτον, η συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης δίνει κίνητρο στην Ελλάδα να επιτύχει επενδυτική διαβάθμιση στα ομόλογα του δημοσίου για να επωφεληθεί έστω με καθυστέρηση πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος γρήγορα. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Ευχαριστώ. Το πρώτο έχει να κάνει με το απόθεμα. Το βασικό εδώ πέρα είναι ότι διατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά που υπάρχουν και τώρα. Και ήταν σημαντική η πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και προερχόμενη από μια κατάσταση που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη, για να μην πω τίποτα άλλο, η Ελλάδα διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη σχετικά. Και το βασικό είναι να διατηρηθεί αξιοπιστία από την οποία χαίρει η Ελλάδα σήμερα. Οι Ιδιαίτερε ευρωπαϊκέ συνθήκες όσον αφορά δηλαδή ε, την κεφαλαία αγορά. Οπότε το βασικό στοιχείο είναι αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του κανείς για την δημοσιονομική πολιτική. Τα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τους στόχους, όχι μόνο μία φορά μάλιστα, παραπάνω. Οπότε συνολικά οι οικονομικές εξελίξεις αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τώρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η μείωσή τους παραμένει ζωτική σημασίας. Και αυτό γιατί με το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι που δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά και αλλού όπου είναι μεγάλο το, ο μεγάλος αριθμός των δανείων αυτών, οδηγούν σε ε, ευπάθεια το τραπεζικό σύστημα. Ε, το οποίο έτσι δεν χρηματοδοτεί επαρκώς τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε είναι προ το συμφέρον τη χώρα να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς βέβαια να πληγεί η συνήθεια, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές και να μην πληγεί η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέου. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το βάρος που έρχεται με τα δάνεια αυτά. Όχι, αλλά είναι δύο πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωριστά. Δηλαδή να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση των δανείων αυτών, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική πτυχή, τις δημοσιονομικές πτυχές. Αλλά είχατε και μια τρίτη ερώτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι ακριβώς ρωτήσατε. Είπα ότι είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν συμμετείχε. Α, ναι. Ξέρετε ότι αυτό έχει να κάνει με την επιλεξιμότητα. Και πιστεύω ότι όταν τα πράγματα συνεχιστούν όπως πάνε μέχρι τώρα και αν συνεχιστεί αυτή η σημαντική πρόοδος της μεταρρυθμίσεις, τότε θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις και θα μπορέσει να συμμετάσχει στην ποσοτική χαλάρωση και η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Πολ Τάνκ. Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε κύριε Ντράγκη, κύριε πρόεδρε της ΕΚΤ. Είναι η τελευταία φορά και τις τελευταίες εβδομάδες κάνατε και πολλούς εχθρούς. Δεν έχετε λόγο τώρα να είστε επιφυλακτικός, δώστε το. Ε, πέστε την γνώμη σας όπως θέλετε. Ε, για την Ολλανδία είπατε ότι έχει 50 δις η Ολλανδία έχει 50 δις για επενδύσεις και του είπατε γιατί δεν τα επενδύει η Ολλανδία. Λοιπόν, από την αρχή το πάω πάλι. Στην συνέντευξή σας, ε, συνέντευξη τύπου πριν από 1,5 μήνα, ε, πήρατε το παράδειγμα της ε, Ολλανδίας και είπατε ότι η Ολλανδία έχει όλα αυτά τα δις ε, και δεν τα επενδύει. Αν τελικά η Ολλανδία δεν το κάνει, θα νιώσετε απογοητευμένος. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, είδα μία εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας που λέει ότι στις μακροπροληπτικές μας εκτιμήσεις θα μπορούσαμε να λιάνουμε ακόμα περισσότερο τον επιχειρηματικό κύκλο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία διατίθενται με χαμηλά επιτόκια και μια νομισματική πολιτική η οποία οδηγεί στην ευελιξία. Εσείς δεν πιστεύετε ότι με την πίεση της ε, ΕΚΤ, μάλλον ότι αρκεί αυτή η πίεση από την ΕΚΤ, η μακροπροληπτική πολιτική λειτουργεί σωστά, με άλλα λόγια, μήπως θα έπρεπε να έχουμε καλύτερο συντονισμό της ε, μακροοικονομ... μακροπροληπτικής ε, πολιτικής. Δέστε λιγάκι τα αρνητικά επιτόκια. Βλέπουμε αυξάνεται ο τομέας της στέγασης, αλλά έχουμε και χώρες οι οποίες δεν έχουν αποθέματα αντικυκλικά, ε, δεν μειώνονται οι τιμές στέγασης. Εγώ ως πολιτικός ανησυχώ που βλέπουμε κάποιες αγορές να ανθούν, αυτό όμως φοβάμαι ότι δεν οδηγεί σε μια ευημερούσα οικονομία. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, νομίζω ότι ο δρόμος προς τα είναι η δημοσιονομική πολιτική αποτελεσματικό συμπλήρωμα της νομισματικής πολιτικής και να είναι αποτελεσματικός μακροοικονομικός σταθοποιητής, αυτός ο δρόμος είναι ένας μακρύς δρόμος και πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν απογοητεύομαι από ένα και μόνο γεγονός, είναι ένας μακρύς και ε, δύσκολος δρόμος. Τώρα είμαστε όμως σε μια κατάσταση συνδυτοποίησης και είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν από δύο ή τρία χρόνια. Είναι μια σταδιακή διαδικασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι τις εξελίξεις ε, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, να επισημαίνουμε το τι πρέπει να γίνει. Το δεύτερο που θέλω να πω φορά στους free rider. Με άλλα λόγια, δηλαδή η ΕΚΤ έχει αρκετή εξουσία για να εμποδίσει χώρες να ξεφεύγουν από την υποχρέωση να εφαρμόζουν μακροπροληπτικά εργαλεία. Κοιτάξτε, ε, όταν συστήθηκε η ΕΚΤ αυτό δεν ήταν ε, μία απόφαση που να λέει ότι θα είναι μία, ε, ένας φορέας ε, που θα εφαρμόζει πολιτική. Θα είναι περισσότερο συμβουλευτικός φορέας που θα εκφράσει τη γνώμη του με συστάσεις και προειδοποίησεις. Τώρα, αν δείτε την εμπειρία μας σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, τότε δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου μακροπροληπτικά εργαλεία στην Ευρώπη. Η ΕΚΤ, λοιπόν, έχει Βεβαίως και είμαστε λιγάκι επηρεασμένοι, δεν είμαστε αντικειμενικοί παρεδιωτές, αλλά αυτό που βλέπουμε έχει πολύ θετική επιρροή στη δημιουργία ε, μιας εργαλειοθήκης, στη διεύρυνση της εργαλειοθήκης, έτσι ώστε η μακροπροληπτική πολιτική να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ε, πολύ συχνά ε, αυτές οι μακροπροληπτικές πολιτικές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν πολιτικά και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες ε, που καθυστερούν ή διαφωνούν στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Τώρα, όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, προφανώς είμαστε κάτω από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και έχουμε τη δυνατότητα εποπτεία σε τομεί, όπως είναι ε, το μέσο των ακινήτων, αλλά αν δεν υπήρχαν τράπεζες, το πρόβλημα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Ε, τους χάρη, ε, οι τράπεζες που δεν είναι παρόντες στον ε, πρωτογενή τομέα του, των ακινήτων, εκεί δεν υπάρχει κανένα εργαλείο η πρόοδος που σημειώνεται στο να ε, δώσουμε στις Εθνικές Αρχές ή στην ΕΚΤ ένα ε, μακροπροληπτικό πλωστάσιο για να μπορούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους στον μη τραπεζικό τομέα, αυτός, ε, αυτές, αυτό ήταν μηδενικό. Και εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα επόμενα έτη. Θα ήθελα ε, να τους, ε, να πω στους συναδέλφους να είναι, ε, να είναι σύντομοι γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ για να μας απαντήσετε για συστημικούς κινδύνους. Επιτρέψτε μου να στρέψω το ενδιαφέρον σας στον τομέα της στέγασης. Το 2018 οι τιμέ ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν πάρα πολύ, κυρίω των σπιτιών, πολύ πιο πάνω από τον πληθωρισμό. Στην Ισπανία κατά 5,1%, στην Ολλανδία κατά 7,4%, στην Πορτογαλία η αύξηση τη κατοικία κατά 9 περίπου%. Ε, στη δική μου την πατρίδα, τη Γερμανία, 5,2%. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση προς εσάς. Ε, υπάρχει κίνδυνος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προκύψει μία φούσκα κατοικίας και ε, με αυτή την πολιτική των μηδενικών επιτοκίων θα ε, παροτρινθούν Ευρωπαίοι να αγοράσουν κατοικία. Και η τρίτη ερώτηση είναι οι τιμές των ακινήτων εκπροσωπούνται στον δίκτυο κατανάλωση έμεσα. Μήπως θα έπρεπε να εκπροσωπούνται άμεσα. Κάνω και την απάντηση. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε συστάσεις. Μισό λεπτό να το δω, γιατί εγώ νομίζω ότι είπα στην εισαγωγή μου ότι έχουμε εκδώσει προειδοποιήσεις προ Γερμανία, Γαλλία, Ισλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία. Όλοι αυτοί έχουν πάρει ε, προειδοποίηση ε, από μας ε, και τώρα έχουν λαμβάνουν συστάσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσουν τις ε, πηγές του ε, συστημικού κινδύνου. Άρα δηλαδή η ΕΚΤ έχει κάνει τη δουλειά της όσον αφορά αυτά τα θέματα. Και ε, αυτό προέρχεται από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Κοιτάξτε, τα αρνητικά επιτόκια σαφώς και παροτρύνουν τους ενδιαφερόμενους να αγοράσουν σπίτια Υπάρχει λοιπόν ε, κάποια δυνατότητα ή είναι αυτό ο σωστό τρόπο για να αλλάξει η νομισματική πολιτική. Ναι, ναι. Η νομισματική πολιτική έχει κατά κύριο λόγο στόχο την σταθερότητα των τιμών και ένας καλός τρόπος είναι να εφαρμόζεται η σωστή μακροπροληπτική πολιτική. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι για το τι θεωρούμε σημαντικό όταν αξιολογούμε ε, την κατάσταση στον τομέα των ακινήτων. Πρώτα απ' όλα, ε, υπάρχουν διαφοροποίηση, μάλλον αξιολόγηση. Αξιολόγηση τα ιστορικά, ε, τους ιστορικούς μέσους όρους, κοιτάμε αν οι αξιολογήσεις είναι τοπικές, ε, αν υπάρχουν κύκλοι, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνουμε την αξιολόγηση. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό σε ορισμένε χώρε, περιορισμό στην προσφορά για πολλού λόγους, ε, περιβαλλοντικούς, ε, σχεδιασμού. Το τρίτο, ε, κατά τον σχεδιασμό των μακροπροληπτικών πολιτικών θα πρέπει κανείς να εξετάζει και την συγκέντρωση των δανειστών ε, σε κάποιους τομείς, ε, το κατά πόσον εκεί ε, υπάρχουν κάποιοι εξαναγκασμοί ε, ή οι οριμάνσεις ε, των υποθηκών, οι βραχυπρόθεσμες υποθήκες μέσα σε 4-5 χρόνια, αυτοί όλοι είναι πιο εκτεθειμένοι στις αλλαγές στις τιμές της κατοικίας, πολύ περισσότερο από ότι σε άλλες χώρες όπου έχουμε σταθερά επιτόκια με μακρύ χρόνο ορίμανσης. Έχουμε μακροπολιτικά μέτρα και για τους δανειστές και για τους δανειζόμενους. Σε κάποιες χώρες ε, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν μέτρα, κυρίως μέτρα για τους ε, δανειζόμενους. Ευχαριστούμε. Κάτω, μέρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τελευταία μου ευκαιρία, κύριε Δράκη, να σας ρωτήσω κάτι που πολλές φορές έχω ρωτήσει και είναι επιπτώσει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημα όμω σήμερα, ακριβώς γιατί εδώ συμπίπτει η συνεδρίαση αυτή με την έναρξη της έσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα. Το 2016 ετοίμασε μια έκθεση η ΕΚΤ που έλεγε ε, πολύ αργά και πολύ λίγα. Εγώ Ξέρω ότι υπάρχει και νέα έκθεση έκτοτε και εκείνη η έκθεση το 2016 ανεφερόταν σε ένα αρνητικό σενάριο όσον αφορά ε, τις αλλαγές στην ε, χρήση της ενέργειας ή την εντατική χρήση του άνθρακα. Τώρα, με το πρόγραμμα της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι θέλει την οικολογική μετάβαση, δηλαδή να επικεντρωθεί διαφορετικά η οικονομία μας ε, απομακρυνόμενη από τον άνθρακα. Αυτά, όπως ε, λέει και η έκθεση, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετική τιμολόγηση της ενέργειας. Οπότε επειδή επήγει το θέμα, τώρα εξαιτία των ε, κλιματικών αλλαγών, μπορώ να σας ρωτήσω πόσο πιστεύετε ε, σοβαρή είναι η κίνδυνη στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα στέλνατε μια προειδοποίηση για το ενεργητικό που συνδέεται με τον άνθρακα ή θα συστήνατε στις τράπεζες να κάνουν κάποιες δοκιμές αντοχής που έχουν να κάνουν ε, με τον άνθρακα, δηλαδή με την έκθεσή τους ε, στον άνθρακα. Απάντηση, όπως σωστά λέτε, όντως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στιμικού Κινδύνου ετοίμασε μια τέτοια έκθεση και εγώ ρώτησα μήπως θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη μια αντίστοιχη έκθεση για το ίδιο θέμα από την Τεχνική Επιτροπή. Έκτοτε από το 2016 δηλαδή οι κίνδυνοι έχουν γίνει περισσότερο ορατοί και περισσότερο εξέχοντες, γιατί όλοι πια τους έχουμε στο μυαλό μας. Η ΕΚΤ εργάζεται με διάφορες ομάδες που δρούν στο τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε πράγματι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα μπορούσε να ετοιμάσει σύντομα και ένα έκθεση. Η κλιματική αλλαγή επίσης είναι κάτι που εξετάζει και η ΕΚΤ και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Η ΕΚΤ, για παράδειγμα, κάνει διάφορα πράγματα επ' αυτού. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό, έτσι δεν είναι. Που είπαμε για τα συνταξιδοτικά ταμεία, για παράδειγμα, που έχουν αυτό το κριτήριο, το περιβαλλοντικό. Το βασικό πάντως είναι ότι κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένας γενικός προβληματισμός πώς να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ο ενιαίο παπτικό μηχανισμό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και πιστεύω ότι αυτό ο γενικό προβληματισμό θα οδηγήσει σε περισσότερο ενεργό και παρούσα συμμετοχή των τριών αυτών οργάνων στον τομέα αυτών. Και πιστεύω την έχω ακούσει, η διάδοχός μου θα δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο ίδιο αυτό μέτωπο. Ευχαριστούμε Φραντσέσκα Ντονάτο από την ομάδα ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως προς τον συστημικό κίνδυνο ήθελα να επισημάνω το εξής. Την κατάσταση που επικρατεί στην Deutsche Bank, τη γερμανική τράπεζα. Ξέρουμε ότι η χρηματοοικονομική της κατάσταση είναι δυσχερής και ξέρουμε ότι κατέρευσε και το σχέδιο συγχώνευσης με την Commerzbank, την άλλη γερμανική τράπεζα. Κατά την άποψη πολλών παρατηρητών, λοιπόν, υπάρχουν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε πτώχευση. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, Πρόεδρε Ντράγκη, το εξή. Κατά την άποψή σας, εάν η Deutsche Bank φτάσει σε πτώχευση, θα πρέπει να εφαρμοστεί μάλλον η νομοθεσία περί διάσωσης, περί bail-in, εξαγοράς. Αλλά αυτό θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις χρηματοοικονομικές και οικονομικές για το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Και λογικό είναι να υποθέσει κανείς ότι για αυτό το λόγο η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τα του bail-in, αλλά να δώσει την έναρξη του bail-out, της εξαγοράς. Αυτό λοιπόν, τι μας δείχνει το σύστημα του Μπέιλιν και η, η όλη ε, σχετική νομοθεσία πως χάσει την αξιοπιστία της όταν έχουμε φαινόμενα αυτού του είδους. Και κατά δεύτερον, επειδή η Deutsche Bank, όπως και άλλες της Βόρειας Ευρώπης, του Βορρά μάλλον της Ευρώπης, έχουν συλλογισμό με πολλά περίπλοκα παράγωγα και αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία κριτική κατά των τραπεζών αυτών. Δεν το σύστημα εποπτεία και παρακολούθηση δεν θα πρέπει να ε, επικεντρώνεται και σε αυτά τα σημεία, αντί να ασχολείται και με, την, ε, με τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μόνο. Διότι αυτοί οι συλλογισμοί που είναι τόσο σύνθετοι και ε, ευπαθεί μπορεί να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμα συστημικό κίνδυνο. Ευχαριστώ. Αν δεν σα πειράζει, θα απαντήσω αγγλικά. Κατά πρώτον, δεν συζητάμε με μονομένα ιδρύματα. Και μετά οι κανόνες του bail-in ή του bail-out είναι κανόνες που ισχύουν κανονικά για όλες τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο. Είναι κανόνες της οδηγίας BRD και από το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τον Ενιό μηχανισμό διάσωσης. Αφορούν όλες τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο. Και ταυτόχρονα Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν και τα στοιχεία του ενεργητικού επίπεδου 2 και 3, όπως τα λέμε. Σε μερικές τράπεζες υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Αλλά διχάνουν χάνουν τις ίδιες προσοχές που έχουν λάβει και τα μη εξυπηρετούμενα διαδάνεια, τα NPL. Και στην έκθεση της ΕΚΤΑ από το Δεκέμβριο θα μπορούσατε να το δείτε. Αλλά και το σκέλος εποπτείας της ΕΚΤ έχει σχολιάσει το σημείο αυτό και μάλιστα περισσότερο επικριτικά από στο παρελθόν τα τελευταία τρία χρόνια. Η διαδικασία λοιπόν έχει ήδη εκκινηθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαν Όβαρτφελτ, ECR. Κύριε Ντράγκη, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι εξελίξεις των τομέα των ακινήτων είναι πολύ σημαντικές γιατί όπως βλέπουμε την τελευταία δεκαετία μια τέτοια είδου κρίση ε, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη οικονομική ε, κατάρρευση το θέμα των επιτοκίων της ΕΚΤ, αυτό έχουμε αφενός και από την άλλη βλέπουμε ότι επιμένεται να υπάρχουν πιο αυστηρές ρυθμιστικές πολιτικές. Αυτό είναι μια παρατήρησή μου. Σχετικά με την ε, χρηματοψηφιακή σταθερότητα βλέπουμε ότι τα φάντα και οι ασφαλιστικές εταιρείε περνάνε δύσκολα ε, διότι τα επιτόκια που εφαρμόζονται είναι πολύ χαμηλά και αυτό υπονομεύει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα ήθελα να έχω τα σχόλιά σας ε, για κάποιες αναλύσεις που έγιναν πρόσφατα ε, σχετικά με τα, τις εγγυήσει και τα παράγωγα. Αυτά μας ανησυχούν λιγάκι. Ε, θα θέλαμε να έχουμε την άποψή σας επ' Σωστά είπατε. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στις χειρότερα μακροπροληπτικά εργαλεία ε, και πολιτική αρνητικών επιτοκίων. Το δεύτερο αφορά το σύνολο της μακροοικονομικής κατάστασης. Το πρώτο είναι περισσότερο εμβαλωματικό και αφορά ε, ε, κάποιες συγκεκριμένες αγορές, αλλά τα δύο αυτά συμπληρώνονται και δεν βρίσκονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Ε, χάρη λοιπόν στην δύναμη, στην ισχύ του μακροπροληπτικού ε, και του μικροπροληπτικού πλαισίου και του ρυθμιστικού πλαισίου, ε, χάρη αυτών η νομισματική πολιτική μπορεί να είναι τόσο εύκολη και τόσο επεκτατική. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τα συνταξιωτικά ταμεία. επ' αυτού οι κίνδυνοι για τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι σημαντικοί ε, για όσους ε, προσφέρουν συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες εδώ ένα σημαντικό εργαλείο είναι η ρευστότητα και οι ιδιωτικέ επενδύσεις ε, ίσως ε, να αντιμετωπίσουν περισσότερους κινδύνους. Μία μακροοικονομική πολιτική θα πρέπει λοιπόν να καλύπτει και τον ιδιωτικό συνταξιδιωτικό τομέα. Η επέκταση όμως ε, των δημοσίων συντάξεων αφορά ένα σημαντικό ποσό των δημόσιων δαπανών και υπάρχουν δημογραφικές ε, προκλήσεις. Αυτά όσον αφορά τα συνταξιωτικά ταμεία. Αλλά είναι σαφώς ε, σωστό ότι η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η δημιουργεί δυσκολίες στα συνταξιωτικά ταμεία και σε λιγότερο βαθμό στις ίδιες τις συντάξεις, αλλά πράγματι δημιουργεί προβλήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, όσον αφορά τώρα δανεισμό με εγγύησης. Το που βλέπουμε σήμερα, ε, κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείες, είναι ότι υπάρξει, υπάρχει υποβάθμιση της αξίας των αγγίσεων που πρέπει να υφίστανται για να μπορεί να χορηγηθεί δανεισμός. Και αυτό Βεβαίως υπάρχει κατά κύριο λόγο στις τράπεζες, αλλά πολύ περισσότερο ε, εκτός τραπεζικού τομέα. Άρα δηλαδή αυτά είναι λιγότερο, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σοβαρά, ε, απλά έχουμε λιγότερα εργαλεία και δεν είναι όλα αυτά τόσο ορατά. Χωσέ Γκουσμάο από την ΚΟΕ. Θα τα πω πορτογαλικά. Ένας από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που έχει εντοπιστεί έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι βιώσιμα κάποια δημόσια χρέη, αλλά και κάποια ιδιωτικά. Πώς εκτιμά, εκτιμάτε εσείς και το Συμβούλιο σας το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τους μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν προκύψει λόγω της, ε, της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Διότι αν αυτές οι ανισορροπίες παραμείνουν στην Ευρωζώνη, στις οικονομίες με μεγάλα ελλείμματα και υψηλό χρέος θα υπάρχει ένα πρόβλημα από άποψη λογιστικής καταγραφής που θα μπορεί να επιληθεί μόνο με πολιτικές συνοχής για να καταπολεμήσουμε ακριβώς αυτές τις ανισορροπίες, τέλος πάντων ελλείψεις ισορροπίας. φαίνεται να περνάμε σε αδιέξοδο. Αν λέμε ότι οι οικονομίες που έχουν πρόβλημα ελλείμματο, επειδή είναι υπερχρεωμένε, δεν μπορούν να εκτελέσουν δημοσιονομικές πολιτικές που επιτρέπουν να διορθώσουν τα ε, διορθωτικά τους προβλήματα. Και επίσης δεν μπορούν, και αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας θέσουν, να ξεκινήσουν προγράμματα εξυγίανσης του χρέους. Συγγνώμη, αλλά έχετε χρόνο για μία μόνο ερώτηση. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας για το συνδυασμό, το συσχετισμό μεταξύ αυτών των δύο προβλημάτων. Ευχαριστώ. Συμφωνώ οι αποκλήσει, οι ανισορροπίε, η έλλειψει ισορροπίε γίνονται χειρότερε με το υψηλό επίπεδο χρέου. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο που βάζει την Ευρωζώνη σε καλύτερη θέση από άλλα μέρη του κόσμου. Υπό την έννοια το ιδιωτικά, τα χρέη των ιδιωτών είναι χαμηλότερα από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται, ιδίως μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Όμως είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το παρελθόν. Τα χρέη όμω των ιδιωτών σταδιακά περιορίζονται να σημειώσω ότι αποκλήσεις και ενισορροπίες έχουν ε, μειωθεί στην Ευρωζώνη. Ε, είπα προηγουμένως ότι η, πρόσθε, η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη και ο κατακρεματισμός της έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ ως προς το πόσο χαμηλός είναι. Ε, Βεβαίω από τι επενδύσει μπορεί να υπάρξει αντίκτυπο, αλλά χρειάζονται και διορθωτικέ μεταρρυθμίσει. Είναι καθοριστική σημασία. Ευχαριστούμε. Ντανούτα Χούμπνερ από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω. Η μία έχει να κάνει με τα, νέα, είδη κινδύνου που αναδύονται και που συνδέονται με το περιβάλλον ή με το κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου τους λαμβάνει υπόψη και μετά τις τελευταίες δοκιμές αντοχής που έγιναν από τον ΙΟΠΑ την Αρχή Επαγγελματικών ε, Συντάξεων. Επίσης η ΕΚΤ θα κοιτάξει και το τραπεζικό τομέα και θα σχεδιάσει και ε, δοκιμές αντοχής που να συνδέονται με αυτούς τους νέους κινδύνους. Δεύτερον, του χρόνου νομίζω θα έχουμε την αναθεώρηση ε, της αφαιρεγγιότητας 2 προκειμένου να συμπεριληφθούν θέματα στο κατάλογο που δεν υπάρχουν σήμερα στο μακροπροληπτικό πλαίσιο. Η ΕΚΤ πριν από ένα χρόνο νομίζω πρότεινε διάφορες παρεμβάσεις, προτάσεις τουλάχιστον, που πηγαίνουν πέρα από το διεθνές πλαίσιο. Οπότε η ερώτηση μου είναι, σε μια τέτοια κατάσταση, σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος η ευρωπαϊκή ασφάλιση να βρεθεί με ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Και είναι σωστό αυτό που κάνουμε μερικές φορές, δηλαδή ότι πηγαίνουμε πέρα από τις παγκόσμιες απαιτήσεις. Έχετε κάποιο παράδειγμα για το ότι κάνουμε καλά ή αντίθετα ότι δεν κάναμε καλά. Απάντηση. Στην πρώτη ερώτηση η απάντηση είναι για του κίνδυνου που έχουν να κάνουν με τον κυβερνοχώρο. Τους συστημικούς κινδύνους που έχουν να κάνουν με τον κυβερνοχώρο. Το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Πρώτα απ' όλα το Γενικό Συμβούλιο καθόρισε ε, και δημιούργησε μία ομάδα που εξετάζει ακριβώς τον συστημικό κίνδυνο στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ευπάθειες και επίσης έχει προβεί και σε μία ανάλυση σεναρίου με αναλυτικό πλαίσιο για να κατανοήσουμε πώς θα ε, δημιουργώντα συστημικός κίνδυνος από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και έτσι ε, θα έχουμε στα τέλη της χρονιάς μια έκθεση που θα αναφέρεται ακριβώς αυτό. Τώρα, είναι σαφές ότι για να γίνει συστημική μια επίθεση στο κυβερνοχώρο θα πρέπει να πλήξει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Πέρα από κάποιες επιτόπου δυσκολίες. Τώρα έρχομαι στο θέμα της ασφάλισης. Σίγουρα επηρεάζεται και ο κλάδος των ασφαλίσεων από την κλιματική αλλαγή ε, και από τις δύο πλευρές του ισολογισμού όσον αφορά το ενεργητικό εξαιτία του μεταβατικού στοιχείου και από πλευράς ε, του παθητικού μπορεί να υπάρξει αύξηση ε, στις απαιτήσει σε σχέση με τώρα. Όλες αυτές τις πλευρές πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και κυρίως ε, βέβαια η αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Εννοείται ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η αντοχή του κλάδου. Τώρα για τη φερικιότητα 2 με ρωτάτε κατά πόσο η θέση σε εφαρμογή της θα βάλει τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες σε θέση ανταγωνιστικού μειονεκτήματος παγκοσμίω. Δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο υπήρξε εντατικός διάλογος ανάμεσα στις επιχειρήσεις ασφαλίσεων και μας εδώ και αρκετά χρόνια. Τέλος, Αφρισάντ, ε, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, το Συμβούλιο Συστημικού κινδύνου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, θα ήθελα να έχω κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το πώς ε, το Συμβούλιο εξετάζει τις ε, μικρομεσαίες τράπεζες, κυρίως τις μικρότερες χώρες. Οι τράπεζες αυτές καλύπτουν κάποια κενά και ε, κενά που προκύπτουν από μεγαλύτερους φορείς. Ε, αυτά τα κενά είναι πολύ μικρά για να τραβήξουν, να προσελκύσουν τις μεγάλες τράπεζες, εκτός αν υπάρξει μια πολύ μεγάλη συμφωνία όλα αυτά φαίνεται ότι αυτές οι μικρότερες τράπεζες, μερικές εκ των οποίων θεωρούνται συστημικές, αυτές επιβαρύνονται με νέα ε, ρυθμιστικά μέτρα. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα, αλλά ε, όμως αυτά τα μέτρα ε, ενισχύουν το λειτουργικό κόστος των τραπεζών και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις νεοφύης επιχειρήσεις. Οι τράπεζες ε, τελικά δεν εφαρμόζουν νέα προγράμματα και πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν έχουν καμία δυνατότητα δανεισμού. Μήπως μπορεί να κάνει κάτι ε, το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο ε, πρόβλημα των μικρών τραπεζών που έχουν να αντιμετωπίσουν κανόνες που είναι απλά γενικευμένοι, έτσι ώστε να ισχύουν για όλους. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας αφορά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο Δηλαδή, αν δείτε λιγάκι το τραπεζικό σύστημα σήμερα στην Ευρωζώνη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι ότι υπάρχει υπερβολικός αριθμός τραπεζών. Έχουμε μείγμα θεσμών, μικρές, μεγάλες τράπεζες, ε, με πολλές και διαφορετικές ε, διαρθρωτικές αδυναμίες, διαφορετική ευαισθησία. Δεν υπάρχει αυτή η συνταγή ε, γενικευμένο να ισχύει για όλους. Παράλληλα υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές τράπεζες. Νομίζω μία παραμφερής ερώτηση που ετέθηκε προηγουμένως το κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει αρνητικά ε, τη δυνατότητα δανεισμού των ε, μικρών ε, τραπεζών. Κοιτάξτε, μικρές και μεγάλες τράπεζες έχουν διαρτρωτικές αδυναμίες και παράλληλα υπάγονται και στους ίδιους κανόνες. Έτσι λοιπόν από τη μια πλευρά θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, προσαρμοστικότητα στους κανόνες, έχοντας κατά νου ότι κάποιοι κανόνες συνεπάγονται την ε, γραφειοκρατική, ε, τήρηση κανόνων ε, από πλευράς μικρών τραπεζών, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Ε, από την άλλη γίνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Βεβαίως και μπορούν να γίνουν περισσότερα, αλλά όσο έχουν τώρα τα πράγματα δεν προβλέπεται διαχωρισμός ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες τράπεζες. Παράλληλα κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες προκύπτουν ακριβώς γιατί είναι μικρές οι τράπεζες. Αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ως εκ τούτου η διαδικασία διαδικασία θα πρέπει ε, να προχωράει ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντράγκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. I like this. Okay. No, I'm not throwing. Okay. Όχι, δεν πρόκειται να σας πετάξω το σφυρί. Απλώς αναρωτιόμουν ε, γιατί υπάρχει. Αλλά να, τώρα κατάλαβα που χρειάζεται. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε αλλά περιμένουμε πρώτα να καθίσουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Προηγουμένως θα σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι συστάσεις και αποφάσεις της 18 ε, και 27 Ιουλίου από πλευράς των συντονιστών. Πώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που ξεκίνησαν στην προηγούμενη θητεία. Επ' αυτού αποφασίσαμε για τους φακέλους που έχουν να κάνουν με τη συναπόφαση ότι ήδη έχουν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση διάφοροι φάκελοι και όσοι είχαν ήδη οριστεί συγκητές και όλες παραμένουν. Για, τους, ε, για τις θέσεις για τις οποίες δεν έχει επανεκλεγεί ο Ευρωβουλευτής ε, θα αναλάβουν νέα από την ίδια πολιτική ομάδα. Τώρα για τις άλλες ε, περιπτώσεις στο κάθε φάκελο συνεχίζουμε από εκεί όπου είχαμε σταματήσει με εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές που έχουν επανεκλεγεί να παραμένουν υπεύθυνοι για το φάκελο. Άλλοι βουλευτές από την ίδια πολιτική ομάδα όμως αντικαθεστούν εκείνους που δεν έχουν επανεκλεγεί. Ε, πρόκειται για τους εξή φακέλους. Πρώτα απ' όλα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οδηγία. Οι συντονιστές ε, συμφώνησαν με την απόφαση των προηγούμενων συντονιστών να χωριστεί ο φάκελος και να υπάρξει νέα προθεσμία για τροπολογίες. Όσον αφορά το ΕΝΤΙΣ, συμφωνήθηκε νέα προθεσμία για τροπολογίες να οριστεί Έπειτα όσον αφορά τις στατιστικές για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, ε, συμφωνήθηκε για το φάκελο αυτό, ο οποίος είχε μείνει αδρανής για πολύ καιρό, να μην αφήσουμε να εκπνεύσουν οι προθεσμίες. Έπειτα για το EISF και το RSP, ε, θέλουμε νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, οπότε θα τεθούν νέες προθεσμίες για τροπολογίες. Επίσης για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ε, αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών. Για τους άλλους φακέλους αποφασίστηκε ότι η ΕΚΟΝ θα ζητήσει από την διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει ότι η Επιτροπή μας θα συνεχίσει το έργο της για άλλους φακέλους χωρίς να πούμε τίποτα πιο συγκεκριμένο. Ορισμοί. Ε, Πωλήσει εξ ε, θα το πάρει ομάδα Renew. Απαιτήσει για υπηρεσίε πληρωμών, το ΕΛΚΑ. Μέτρα για ενίσχυση διοικητική διαδικασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απάτε των ΦΠΑ, ΕΛΚΑ. Πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2006-112 ΙΣΥ όσον αφορά το κοινό σύστημα ε, ΦΠΑ και την Οδηγία 2008-118 ΙΣΥ σχετικά με τις γενικές διευθετήσεις για τους φόρους πολυτελείας οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευρωπαϊκό εξάμεινο για το συντονισμό οικονομικών πολιτικών, οικονομικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ, ΕΛΚΑ βεβαιώνεται. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ετήσια έκθεση, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, πολιτική ανταγωνισμού, ετήσια έκθεση, το Ρινιού. Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Γενικός προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό του 2020, όλα τα τμήματα, ΕΛΚΑ οι οικονομικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσουν ετήσια έκθεση ή πράσινη τον αλαμβάνουν. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι συντονιστέ επιβεβαίωσαν το χρονοδιάγραμμα τη ΕΚΟΝ μέχρι τα τέλη του 2019 και συμφώνησαν για ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τι συνεδριάσει μα το 2020. Επίση, οι συντονιστέ συμφώνησαν για χρονοδιάγραμμα συναντήσεων συντονιστών μέχρι τα τέλη τη χρονιά αυτή. Ε, αποστολή μας στην ετήσια συνάντηση στην Ουάσιγκτον του Διεθνούς Μασματικού Ταμείου, 16 με 20 Οκτωβρίου. Συμφωνήθηκε ότι σύμφωνα με το σύστημα DONT θα καθοριστεί η σύσταση, δύο από το ΕΛΚ, δύο από τους ουσιαστέ και Δημοκράτες, ένας από το ΡΙΝΙΟΥ, ένας από τους Πράσινους και ένας από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Τέλος, συμφωνήθηκε να οργανωθεί ακρόαση στην ΕΚΟΝ στις 5 Σεπτεμβρίου με την Επίτροπο Γιούροβα και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Κάμπα όσον αφορά την εφαρμογή του AMLD, δηλαδή Οδηγία για ε, πρόληψη νομοποίησης εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Θα προσκληθούν και οι ΛΥΜΠΕ. Αλλά βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει αφού αφορά την 5η Σεπτεμβρίου. Και συμφωνήθηκε να προσκαλέσουμε και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνάντηση της ΕΚΟΝ πριν από τα τέλη της χρονιάς. Αυτό όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια δοκιμή για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ο κύριος Κίρτσος δεν έχει μαζί του την κάρτα του. Θα προσθεθεί στο αποτέλεσμα η ψήφος του. Ωραία, τελειώσαμε και με το τεστ. Πρώτη ψηφοφορία. πρόταση για κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ε, παρόχους υπηρεσιών crowdfunding για επιχειρήσεις. Απόφαση για να περάσουμε σε διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. 33 υπέρ 12 κατά 34 με μία πρόσθετη 12 εγκρίνεται και επόμενη πρόταση για κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2014-65 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αγορές χρηματοοικονομικών εργαλείων. Απόφαση και πάλι για να περάσουμε σε διαθεσμικές δια... διαπραγματεύσεις. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Δεν ψήφισαν άπαντες. Ωραία, πέρας. 34 συν 1 υπέρ, 12 κατά, καμία εποχή εγκρίνεται. Okay, so this meeting is finished. Κυρίσω την λήξη της συνεδρίασης, συνεχίζουμε αύριο στις 2.30. Ευχαριστώ.